Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Να σας παρακαλέσω, όσοι θέλετε να μείνετε μαζί μας, να καθίσετε και να ξεκινήσουμε με το σημείο 17 της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην τρέχουσα κατάσταση και τις μελλοντικέ συνέργειες για αυξημένη αποτελεσματικότητα μεταξύ του ΕΤΠΑ και άλλων διαρθρωτικών ταμείων. Είναι μια έκθεση της πρωτοβουλίας ε, του Γεωργίου Σταυρακάκη και σήμερα θα γίνει ανταλλαγή απόψεων όχι μόνο με τον εισηγητή της έκθεσης αλλά και με προσκεκλημένους ομιλητές. Θα παρουσιάσω τους προσκεκλημένους ε, μετά την ε, εισαγωγή του κυρίου Σταυρακάκη. Ξεκινώ λοιπόν ζητώντας από τον κύριο Σταυρακάκη να παρουσιάσει τα εισαγωγικά του σχόλια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, η κύρια παραδοχή γύρω από την οποία αναπτύσσεται το έγγραφο εργασίας που έχετε στη διάθεσή σας είναι ότι οι ενισχυμένες συνέργειες μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής μπορούν να διασφαλίσουν καλύτερα αποτελέσματα για τη μεγέθυνση και την ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο και μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για την διαθέσιμη χρηματοδότηση από ό,τι το κάθε ταμείο μόνο του. Η ιδέα που περιγράφεται στο έγγραφο είναι ότι για να πετύχουμε πραγματική προστιθέμενη αξία χρειαζόμαστε μια στρατηγική προσέγγιση και κοινού κανόνες εφαρμογής για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο γενικό πλαίσιο της πολιτικής της συνοχής, καθώς και με το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο για την Αγροτική Ανάπτυξη και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλλιές. Γενικότερα, η ανάγκη για συντονισμένη προσέγγιση όχι μόνο για τα μέσα της πολιτικής συνοχής, αλλά και για όλα τα άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως για την έρευνα, την καινοτομία, τη διαβίου μάθηση και τα δίχτυα, αναγνωρίζεται ρητά και από την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση του προπολογισμού όπου προτείνεται ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο προκειμένου να διασφαλιστεί μεγαλύτερος συντονισμός. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεδομένης της στενότητας του χρόνου δεν θα ήθελα να σταθώ σε λεπτομέρειες του εγγράφου εργασίας, εξάλλου το έχετε. Αφού ευχαριστήσω θερμά τους εκλεκτούς προσκεκλημένους μας για τη συμμετοχή τους στη σημερινή συζήτηση, θα ήθελα η κυρία Πρόεδρος να τους δώσει το λόγο προκειμένου να δούμε μέσα από την πολύτιμη εμπειρία τους πρακτικά ζητήματα των θέσεων που αναπτύσσονται στο έγγραφο εργασίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σταυρακάκη. Έχουμε τρεις προσκεκλημένους ομιλητές τον ε, Γιάν ε, Μάρτιν Τεφέτ, διευθυντή του ΕΚΟΡΙ της Βρυξέλλες, μια ε, εταιρεία συμβούλων και έρευνα, τον Χέλερ Νόρμπερτ, διευθυντή της Αρχής Διαχείρισης της Αξονία Άνχολτ στη Γερμανία και τον Σεραφίν Πάζος Βιδάλ, επικεφαλή του γραφείου Κόσλα στις Βρυξέλλες και αυτό είναι μια σύμβαση των τοπικών αρχών της Σκωτία. Καλό πρώτα τον Γιάν Μάρτιν Τεφέτ να λάβει το λόγο. Κύριε Τοφέτα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι καλημέρα. Θα ήθελα να επικεντρώσω την παρέμβασή μου σε, στις εμπειρίες του Ερμαντή από την ε, αξιολόγηση που έκανε η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή σε, για ένα πρόγραμμα ε, στην περίοδο 2001-2006 το οποίο στοιχίζει 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Το πρόγραμμα Urban 2 είναι ένα παράδειγμα μιας ε, ολοκληρωμένης σειράς πολιτικών, όχι μόνο στη θεωρία αλλά και στην πράξη. Και εδώ αναφέρομαι σε μια βασική πρόκληση για όλα τα ταμεία συμπεριλαμβανομένου και του ΕΤΠΑ να επικεντρωθούν στα πραγματικά προβλήματα των ε, πόλεων και των αστικών περιοχών. Έχουμε λοιπόν την εμπειρία του ΕΡΠΑΝΤΟΥ που μας δείχνει πώς γίνεται κάτι τέτοιο. Το πρόγραμμα ε, έτρεξε την περίοδο 2001-2006 και ανέπτυξε αναπτυγμένες και ανανεωμένες ε, προσεγγίσεις για την αναγέννηση των ε, περιοχών και γειτονιών σε κρίση. 7,5 εκατομμύρια ευρώ ήταν τα κονδύλια που δεσμεύτηκαν για τα 14 κράτη-μέλη που συμμετείχαν, τα οποία ε, καλύπταν 2,2 εκατομμύρια ε, κατοίκους συνολικά. Έτσι λοιπόν η ολοκλήρωση των συνεργειών και των ε, πόρων χρησιμοποιήθηκε για να αυξηθεί ο αντίκτυπος με πολλούς τρόπους. Καταρχάς ε, μέσω της ε, ολοκλήρωσης των προγραμμάτων στρατηγικών και πόρων, δεύτερον μέσω της ολοκλήρωσης σε επίπεδο project προγραμμάτων, τρίτον μέσω συνεργειών μεταξύ του προγραμμάτων του Urban και μέσα από ολοκληρωμένες ομάδες εκτέλεσης. Έχουμε τέσσερις τύπους. Πρώτα την ενσωμάτωση των στρατηγικών προγραμμάτων και κονδυλίων. Αυτή η ολοκλήρωση βοηθεί, ε, βοηθά στην ε, κινητοποίηση επιπλέον ε, χρηματοδοτήσεων συμπεριλαμβανομένων και κύριων προγραμμάτων. Τα χρήματα του ΕΤΠΑ, του ΕΡΜΑΝ και άλλων βασικών πόρων ήταν αυτά που ουσιαστικά είχαν το μεγαλύτερο αντίκτυπο και Είχαμε ας πούμε περιπτώσεις όπως ε, την περιοχή Κύχο στην Ισπανία όπου χρησιμοποιήθηκαν τα υπάρχοντα ε, κονδύλια της περιφερειακής κυβέρνησης της Αστούριας ε, για συνδυασμό με τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Δεύτερον, ολοκλήρωση σε επίπεδο προγραμμάτων. Μέσα στα πλαίσια των προγραμμάτων του Urban υπήρξε μεγάλο βαθμό ολοκλήρωση. Ε, πολλά, πολλά προγράμματα στόχευσαν ε, στην πραγματοποίηση και αντιμετώπιση πολλών ε, ε, θεμάτων τα οποία είχαν ως αντίκτυπο κάποια οικονομικά ωφέλη, κάποια κοινωνικά προγράμματα για την απασχόληση των τοπικών γυναικών ή τη φύλαξη των παιδιών κτλ. Στην πόλη του Ρότερνταμ τα κονδύλια χρησιμοποιήθηκαν για μη κοινού σκοπούς δημιουργήθηκε ένα κέντρο νεότητας για μετανάστες και έγινε και ένα project για μια μυστική αποστολή με σκοπό να συλλεχθούν στοιχεία τα οποία θα χρησιμοποιούνταν για να αντιμετωπιστούν τα βασικά προβλήματα αυτής της περιοχής. Έτσι λοιπόν μειώθηκε ε, το έγκλημα στην περιοχή, μειώθηκε ο αριθμός των παιδιών που παρατούσαν το σχολείο και γενικά βελτιώθηκε η κατάσταση. Τρίτος τύπος ε, εναρχίστρωση μεταξύ των προγραμμάτων. Θεωρήσαμε ότι όταν έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να ε, το οποίο θεωρούμε ότι θα λύσει όλα τα ε, κοινωνικά προγράμματα είναι μάλλον αφελές. Ε, υπάρχουν ε, σε περιοχές της Ολλανδίας, για παράδειγμα, τέτοιες προσπάθειες, οι οποίες όμως συμπεριλαμβάνουν μια πλειονότητα προγραμμάτων, εμπειρία από μεγάλες ομάδες, υποστήριξη σε τοπικές επιχειρησιακές ομάδες κτλ το γεγονός ότι αυτά τα προγράμματα αμοιβαία υποστηρίζονται οδήγησε σε μεγαλύτερη πρόοδο και μεγαλύτερο αντίκτυπο. Τέλος, ε, το τελευταίο είδος ε, ολοκλήρωση είναι οι ολοκληρωμένες ομάδες απόδοσης. Σε πολλές ε, περιοχές του Urban χρησιμοποιήθηκε για να δημιουργήσει το περιβάλλον για την ολοκλήρωση των εταιρικών σχέσεων την και την ε, συνεργασία μεταξύ ατόμων ε, σε διάφορες περιφέρειες ε, και φορείς. Έτσι μπορέσαμε να δούμε τη γενική εικόνα, να δούμε ποιες είναι οι συνέργειες που, μας, που διατίθενται Επίσης στο Χάλιφαξ ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο που το Έρμπαν και εθνικά κονδύλια για, από τον τοπικό προπολογισμό αναγέννησης ε, χρηματοδότησαν μια δράση στο Χάλιφαξ. Ε, στη Γαλλία επίσης ε, μια περιφερειακή αρχή υποστηρίχθηκε για να ε, προωθήσει προγράμματα στις νότιες περιοχές της πόλης. Έτσι λοιπόν ο district manager στην περιοχή αυτή κατάφερε να πετύχει πράγματα που δεν θα πετύχαινε με μία αποκλειστικά τομεακή προσέγγιση. Για να καταλήξω λοιπόν να πω ότι το Urban έχει δικαιολογήσει την ε, ύπαρξή του ε, χρειάζεται για να διασφαλίσουμε τον αντίκτυπο ειδικότερα σε περιοχές μετά την κρίση. Και είναι πραγματικά πολύ μεγάλος ο αντίκτυπος αυτός. Το Urban 2 είναι πραγματικά ένα παράδειγμα που μας δείχνει πως μια τοπική ολοκληρωμένη προσέγγιση έχει τόσο καλά αποτελέσματα. Ένα καλό επιχείρημα είναι ότι αυτές οι πολιτικές έχουν πολλές πιθανότητες να ε, μας βοηθήσουν να μην χάσουμε το στόχο από τα μάτια μας. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Νόρμπερτ Χέλης για να μας παρουσιάσει τα σχολιά του. Ε, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω στα γερμανικά. Βλέπετε τη Σαξονία Άνχαλτ στο, μέτρο, στο μέσο αυτής, αυτού του χάρτη. Και εδώ τα περιφερειακά προγράμματα έχουν, ε, καλύπτουν μια μεγάλη επιφάνεια και πρέπει να αναπτυχθούν στρατηγικά σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Ε, όσον αφορά στη συνοχή, γνωρίζετε πολύ καλά τι γίνεται, δεν χρειάζεται να σας τα διαβάσω τι είναι η συνοχή, όμως είναι μια ε, συγκεκριμένη και πολύπλοκη διαδικασία για τις ε, διοικητικές αρχές. Στη δική μας περιοχή ε, είχαμε τρία ταμεία, το περιφερειακό, το έτμα και μια συνολική και το κοινωνικό ταμείο με μια συνολική χρήση 12 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εδώ λοιπόν ε, βλέπετε πως αντιμετωπίσαμε θέματα ε, περιφερειακής ανάπτυξης, ε, είδαμε τι είναι τα σημεία που μπορούν να χρηματοδοτούν, ποιες είναι δηλαδή οι εργασίες που μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε και Είδαμε από τα πολλά προγράμματα Urban ότι το μειονέκτημα ήταν πώς πρέπει, ότι δεν εξηγείται πώς πρέπει να ε, τρέξουν διάφορες διαδικασίες. Υπάρχει λοιπόν, ε, υπήρξε μια στρατηγική προσέγγιση, έγινε μια αξιολόγηση αυτών των διαδικασιών, ε, να μετρήσαμε τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις. Και Τώρα υπάρχει μια διαφορά μεταξύ του αστικού και του μη αστικού περιβάλλοντος ε, όσον αφορά στα σχολεία, στα νηπιαγωγεία, τους δρόμους, ε, τις μικρές επιχειρήσεις, ε, τους βοηθούς νοτομίες, μικρά δάνεια. Όλα αυτά είναι πράγματα που μπορούμε να κάνουμε στο αστικό περιβάλλον αλλά και στο γεωργικό περιβάλλον και είναι κάτι που ενιαία αντιμετωπίζουμε σε όλη την περιφέρεια. Ε, όμως ε, σε επίπεδο τοπικό χρειαζόμαστε διαφορετικές ε, δομές για τις διοικητικές αρχές στην ίδια περιοχή, στην ίδια περιφέρεια. Χρειαζόμαστε κανόνες ε, χρηματοδότησης, επιλεξιμότητας και δυνατότητας χρηματοδότησης κοινέ παρεμβάσεις και κοινή γλώσσα. Χρειαζόμαστε ε, πληροφοριακά συστήματα γιατί ε, τα περιφερειακά, τα διαρθρωτικά ταμεία ε, παίζουν σημαντικό ρόλο όχι μόνο σε επίπεδο θεωρητικό αλλά σε επίπεδο εφαρμογής. Ένα project είτε είναι στην πόλη, είτε είναι στο χωριό, είτε είναι μεγάλο, είτε μικρό είναι πάντοτε ένα πρόγραμμα και σε όλη την Ευρώπη είναι ευρώ που χρησιμοποιούμε. Έτσι λοιπόν πρέπει να δώσουμε κάποιες εξηγήσεις σχετικά με το κάθε πρόγραμμα. Υπάρχουν κάποια τυπικά ε, προγράμματα χρηματοδότησης ε, γεωργικών περιοχών όπως ε, χρηματοδότηση βρώμης κτλ. και άλλα προγράμματα που ενισχύουν την αγορά εργασίας. Απ' την άλλη όμως υπήρχε ένας πυρήνας ο οποίος ήταν κοινό σε όλα τα project και σύντομα ε, είδαμε ότι έπρεπε να δούμε τις ιδιαιτερότητες ε, και να χωρίσουμε τις ομάδες σύμφωνα με αυτές. Έτσι λοιπόν για κάθε project και κάθε αίτηση για project υπάρχει αυτή ως ο κοινό ε, πυρήνας για κάθε ε, χρηματοδότηση, για κάθε αδειοδότηση, για κάθε αξιολόγηση ενός project υπάρχει αυτός ο κοινός ε, πυρήνας. Τι μπορούμε να μάθουμε τώρα από το παρελθόν μας. Χρειαζόμαστε ένα ενιαίο σύστημα διοίκησης για όλα τα ταμεία και για πολλές περιόδους. Το σύστημα αυτό δεν πρέπει να αλλάζει συνεχώς ε, κάθε φορά, δηλαδή που θα αλλάζουμε περίοδο, γιατί μία πέφτει πάνω στην άλλη. Ε, μπορεί να έχουμε τρεις περιόδους που να αλληλοκαλύπτονται. Έτσι λοιπόν, όσοι εργάζονται ε, στα project αυτά στις διάφορες περιφέρειες μπορεί ταυτόχρονα να τρέχουν πολλά προγράμματα τα οποία απαιτούν διαφορετικές διοικητικές προσεγγίσεις και αυτό σε επίπεδο εφαρμογή των ε, προγραμμάτων δημιουργεί σύγχυση. Για να διευκολύνουμε την ε, κατάσταση όταν γίνεται σε κάθε περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα, σε κάθε περιφέρεια. Έχουμε μία ε, αρχή διοικητική, η οποία συζητεί με τις διάφορες αρχές της Βρυξέλλες, την Κομισιόν κτλ. για να μπορεί ενιαία να εφαρμόζεται η διαδικασία και χρειαζόμαστε και τους ίδιους ε, κανόνες ε, χρηματοδότησης ε, για όλα τα ταμεία, ας πούμε, σε επίπεδο ΦΠΑ ή όταν έχουμε το, περιφερειακό, το Ταμείο Κοινωνικής Ανάπτυξης, το οποίο έχει κάποιες φορολογικές απαιτήσεις, ή σε, στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε το ΦΠΑ λοιπά. Όλα αυτά ας πούμε βοηθούν μια επιχείρηση να πάρει πίσω το φόρο από την εφορία της ε, και Υπάρχουν και περιοχές στη Γερμανία, π.χ. που μπορεί να παίρνουν πίσω το φόρο αλλά όχι το ΦΠΑ κτλ. Υπάρχουν αυτές οι διαφορές, αλλά αν έχουμε κοινού ε, κανόνες λύνονται τα προβλήματα. Ένα αρνητικό παράδειγμα είναι κάποια προγράμματα τα οποία είχαν ε, ε, την απέντηση να γίνει επιτόπου έλεγχος ο οποίος έγινε μέσω GPS, μέσω δορυφόρου, για, αφορούσε στην καλλιέργεια κάποιων εδαφών. Και εκεί πραγματικά ε, χρειάζεται μια συγκεκριμένη προσέγγιση, η οποία είναι ε, ιδιαίτερη για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Χρειαζόμαστε τους ίδιους λοιπόν κανόνες αξιολόγησης για, όλους, για όλα τα ταμεία. Ένα άλλο παράδειγμα στο Γεωργικό Ταμείο είναι μια ε, έκθεση ετήσια η οποία ε, απαιτείται είναι μια συνεχής αξιολόγηση και υπάρχει και η στρατηγική αξιολόγηση. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια ενιαία ε, γλώσσα και την ίδια μετάφραση επειδή όλα τα κείμενα πρέπει να χρησιμοποιούν τις ίδιες γλώσσες, τις ίδιες λέξεις, ας πούμε, όταν είναι μετάφραση από τα αγγλικά κτλ. Για παράδειγμα, η... ένα αρνητικό άλλο παράδειγμα είναι οι αρχές που καταβάλουν τις πληρωμές. Ε, επίσης, οι ελεγκτικές αρχές του Αγροτικού Ταμείου πρέπει να διαφοροποιούνται από αυτές των άλλων ταμείων και πολλές φορές υπάρχει σύγχυση γιατί χρησιμοποιείται η ίδια λέξη για την αρχή αυτή. Επίσης είχαμε και προβλήματα με τα καινοτόμα εργαλεία χρηματοδότησης. Η συζήτηση ήταν επιφανειακή και το τι καταλάβαινε κανείς ε, με την κάθε λέξη ε, αλλάζει κατά τη διάρκεια της χρηματοδοτούμενης περίοδου. Δεν υπήρχε λοιπόν πάλι νέα γλώσσα. Στην τελευταία ε, λοιπόν περίοδο μιλήσαμε στη Γερμανία για προεταιρεότητες... το οποίο μεταφράστηκε ως ε, βασικά σημεία. Ε, τώρα πια δεν χρησιμοποιείται αυτή, αυτός ο όρος, αλλά χρησιμοποιείται ο όρος ε, άξονες προτεραιότητας. Έτσι λοιπόν στους κανονισμούς υπάρχουν διαφορετικές λέξεις και υπάρχει αυτή η σύγχυση. Χρειαζόμαστε λοιπόν ενιαίους ορισμούς για όλα τα ταμεία που θα είναι, ισχύουν για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δίνονται κεντρικά από τις Βρυξέλλες για να μπορούμε να κατανοούμε πώς γίνεται ας πούμε, μια πληρωμή η οποία μπορεί να είναι ε, μια προκαταβολή, μπορεί να είναι μια δόση, μπορεί να είναι μια τελική πληρωμή. Επίσης ε, τα λογιστικά στοιχεία είναι ε, σημαντικό να έχουν ενιαία ορολογία. Ε, οι δείκτες ε, στο χώρο εργασίας και πάλι χρειάζονται έναν ενιαίο ορισμό όταν μιλάμε για χώρο εργα... θέσεις εργασίας κτλ. Χρειάζεται λοιπόν ένα πληροφοριακό σύστημα για όλα τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή τουλάχιστον σε επίπεδο κράτους μέλους ή τουλάχιστον σε περιφερειακό επίπεδο. Χρειαζόμαστε ενιαίες επιταγές ε, αξιολόγησης και λογοδότησης γιατί όταν αυτά αλλάζουν ε, είναι δύσκολο ε, κανείς να φτιάξει μια ενιαία τράπεζα πληροφοριών. Χρειάζεται λοιπόν για άλλη μια φορά ενιαία γλώσσα, ενιαίοι ορισμοί, ενιαίες μεταφράσεις και ερμηνείες έτσι ώστε να υπάρχει σύγκριση. Είναι λοιπόν καλύτερα να υπάρχει ένα πληροφοριακό σύστημα μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί να υπάρχουν ε, κατάλληλες ε, πληροφορίες ε, για τη λήψη αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε περιφερειακό, εθνικό και επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να πετύχουμε τον στόχο μας, ε, αλλά όταν έχουμε ταυτόχρονα πολλούς ε, δρόμους δυσκολεύουν τα πράγματα. Θα πρέπει ο καθένας λοιπόν να αποφασίζει από μόνος του ε, πώς, ποια είναι τα προβλήματα επικοινωνίας και να τα δείχνει. Για κοιτάξτε ας πούμε αυτές εδώ τις φωτογραφίες. Στο τέλος θα δείτε, αν κοιτάξετε προσεκτικά τις φωτογραφίες, ποια είναι η διαφορά στο πώς κανείς αντιλαμβάνεται την κούνια. Το παιχνίδι αυτό. Πρέπει λοιπόν ε, να εξετάζουμε την ε, έννοια των όρων ε, για να μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το τι εννοούμε. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank you very much. Was Ευχαριστώ πολύ. Έχει μεγάλη σημασία να ακούμε τους ειδικούς, τους γνώστες για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Και τώρα ο κύριος Βιντάλ ε, Κόσλα από το Γραφείο Βρυξελών των Δήμων. Thank you. Thank you, Chair. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ, ευχαριστώ και τον εισηγητή που μας ε, προσκάλεσε. Είμαι επικεφαλής του γραφείου της τοπικής αυτοδιοίκησης της Βρυξέλλες, αρμόδιος για θέματα συνοχής εδώ και πολλά χρόνια. Είμαι εδώ όμως, κυρίως ως πρόεδρος της ομάδας του CMR για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Πιστεύω ότι καλώς μιλώ τελευταίος μετά από τους ειδικού για τα χρηματοοικονομικά μπορώ να καταθέσω τη γνώμη του ειδικού στη διαχείριση έργων σε τοπικό επίπεδο. Οπότε, ας δούμε την πρώτη διαφάνεια. Καταρχήν, εισαγωγικά, το CMR είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών. Είναι ουσιαστικά η ομοσπονδία όλων των ενώσεων ε, τοπικής αυτοδιοίκησης ανά την Ευρώπη. Είμαστε το αρχαιότερο όργανο στο επίπεδο αυτό. Εδώ και χρόνια, αλλά κυρίως πρόσφατα δουλεύουμε σε θέματα περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης. Είμαστε σύμβουλοι της Κομισιόν, προκειμένου, τα τελευταία δύο χρόνια συγκεκριμένα. Και χαιρόμαστε βεβαίω ε, πολύ που το θέμα αυτό περιλαμβάνεται στην μελλοντική έκθεση, πάνω στην έκθεση για το μέλλον της συνοχής αναζητούμε απαντήσεις σε διάφορα θέματα βάσει όμως των στοιχείων που μας οι ειδικοί και όχι μόνο οι τοπικές μας οι εθνικές ενώσεις. Μιλούμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάνω από 20 χρόνια πείρα στον τομέα και βάσει αυτής της πείρας καταφέρω και τα δικά μας συμπεράσματα. Είμαστε επίση συντονιστές του δικτύου των αεφορικών πόλεων όπως προείπα το Κόσλα είναι μία από τις οργανώσεις μέλη του CMR είμαστε ουσιαστικά μία ένωση τοπικών αρχών στην Σκοτία Οι δήμοι στην περιοχή μας είναι σχετικά μεγάλη με μέσο όρο 162.000 πληθυσμό. Έχουμε πει, όπω είπα, εδώ και πολλά χρόνια στην παροχή συμβουλών και στην διαχείριση έργων για την τοπική ανάπτυξη και αυτοδιοίκηση. Αυτά είναι τα πράγματα, οι πρωτοβουλίε, αν θέλετε, και το οποίο βασίζεται στην εμπειρία που έχουμε συγκεντρώσει τα τελευταία χρόνια. Όπως βλέπετε εδώ, και είναι πράγματα που τα ξέρετε βεβαίω υπάρχουν πολλά και διαφορετικά ταμεία, ίσω περισσότερο και από ό,τι πρέπει λένε ορισμένοι το Περιφερειακό Ταμείο, το Κοινωνικό Ταμείο για τον άξονα 3 ειδικά έχουμε το γενικό Ταμείο το Ταμείο Αλίας και άλλα όπως το δίκτυο για την ευφυή ενέργεια και ούτω καθεξής. Έχουμε ακόμη διαφορετικές πλατφόρμες πάνω στις οποίες μπορεί να στηριχθεί η τοπική ανάπτυξη. Το Urban, για παράδειγμα, το Leader, το Flag στον τομέα της Αλίας. Υπάρχουν λοιπόν δυνατότητες Το θέμα είναι πώς θα ενοποιήσουμε και θα εξορθολογήσουμε όλο αυτό το σύστημα ώστε όλα αυτά να έχουν κάποια προσθεμένη αξία. Επίσης, μας βοήθησε πολύ η εξέλιξη όσον αφορά τα μέτρα γεωργικής ανάπτυξης. Μας βοήθησε επίσης πολύ η συμφωνία του κοινωνικού με το περιφερικό Ταμείο. Αλλά αυτά είναι μόνο η εισαγωγή και η θεωρία. Στην πραγματικότητα, τα πράγματα είναι πιο πολύπλοκα. Μιλάμε καταρχήν για ανθρώπους, ας πούμε ενός μικρού δήμου που μπορεί να έχει μόνο ένα στελέχος, ένα άτομο να ασχολείται με όλα αυτά. Και εντοπίζει μια πολυπλοκότητα. Επίσης, για κάθε ταμείο υπάρχουν διαφορετικές διαχειριστικές αρχές, πολύ συχνά. Υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα διοίκηση και αυτοδιοίκηση που εμπλέκονται. Οι κανόνες τεχάνουν διαφορετικών ερμηνεών πολύ συχνά και αυτό μπορεί να κρίνει την επιτυχία ενός έργου και επιπλέον ακούμε από τα μέλη μας ότι οι διάφορες ερμηνείες ε, από την διαχειριστική αρχή για παράδειγμα δίστανται ή αλλάζουν με το χρόνο. Οι οδηγίε πολλέ φορέ που δίνει η Κομισιόν δεν ταυτίζονται με αυτέ του κράτου μέλου ή δεν φτάνουν στου ενδιαφερόμενου. Και υπάρχουν φυσικά και εθνικέ απαιτήσει οι οποίε ε, είναι και εθνικοί κανόνες βάσει των οποίων πρέπει να γίνει το σχέδιο. Τέλος, Υπάρχουν θέματα χρονοδιαγράμματο, υπάρχουν θέματα τοπικών δυνατοτήτων. Πολλέ φορέ για έναν μικρό Δήμο, ακόμα και ένα μεσαίο Δήμο, είναι δύσκολο, παραλαμβάνω, να διαχειριστεί ένα έργο και όλε αυτέ τι απαιτήσει. Ένα κλασικό παράδειγμα, αν προκειμένου, το οποίο μα επισημαίνουν πολλά μέλη μα, γιατί έχουν σχετική εμπειρία, είναι η υποστήριξη τη αποσχολησιμότητα. Εδώ εμπλέκεται το Κοινωνικό Ταμείο και το Περιφερειακό Ταμείο. το Περιφερειακό Ταμείο ασχολείται περισσότερο με τις γενικές πτυχές. Το κοινωνικό εξειδικεύεται σε προγράμματα που στοχεύουν συγκεκριμένα τύπα του πληθυσμού. Στο τοπικό επίπεδο, τελικώς, μπορεί να υποστηρίζεται το ίδιο άτομο μέσω διαφορετικών μέτρων μέσω του ιδίου ε, στελέχους του Δήμου, αλλά από διαφορετικά ταμεία, κάτι το οποίο δεν έχει πολύ έννοια, όπω καταλαβαίνετε, γιατί μιλάμε για το ίδιο άτομο, το ίδιο πρόβλημα και την ίδια χρονική περίοδο. Ένα άλλο παράδειγμα, το οποίο σημαίνει και αυτό πολύ συχνά, είναι όταν τα δύο αυτά ταμεία μοιράζονται το κόστος για κάποια εγκατάσταση, για κάποια υποδομή. Και εδώ τα πράγματα περιπλέκονται για το πώς θα κατανεμηθεί δηλαδή για παράδειγμα το λειτουργικό κόστος της εγκατάστασης. Υπάρχουν πράγματα που είναι πραγματικά ανατριχιαστικά ε, σε περιοχές ιδιαίτερα όπου οι τοπικές δυνατότητες είναι περιορισμένες. Και υπάρχουν άλλα που ακούγονται αστεία, αλλά δεν είναι. Είναι το λεγόμενο δίλημα του χαρτιού τουαλέτας. Χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο για να περιγράψουμε το εξή πρόβλημα. Όταν αφιερώνουμε πάρα πολύ χρόνο για να κρίνουμε αν κάποια ε, στοιχεία του κόστου, όπως ακόμη και ναι το χαρτί ελέτες ε, πρέπει να καταλογιστεί στο ένα ή στο άλλο ταμείο. Αυτά τα πράγματα αποτελούν γραφειοκρατία που συνεπάγεται καθυστερήσεις βραδείς ελέγχους και επαληθεύσεις και φυσικά όλα αυτά είναι εις βάρος των αποτελεσμάτων. Φυσικά τα δύο ταμεία έχουν μια συμφωνία συγχρηματοδότησης η οποία όμως δεν χρησιμοποιείται πολύ συχνά λόγω της νομικής ασάφειας που υπάρχει όπως καταλαβαίνετε. Άρα το μέτρο αυτό χρησιμοποιείται μόνο σε εξαιρετικέ περιπτώσει. Ιδανικά βεβαίω θα έπρεπε να έχουμε ένα ενιαίο ταμείο. Εν πάση περιπτώσει ε, όλα αυτά καθυστερούν και ε, του ελέγχου και τι επαληθεύσει στο τέλο του καθέργου. Έχουμε ένα άλλο πρόβλημα τώρα. Ένα κατακόρυφο πρόβλημα που αφορά αρμοδιότητες και το σε ποιο επίπεδο εμπλέκονται πλέον οι εθνικές αρχές. Είτε μιλάμε για τη Γαλλία, είτε για τη Γερμανία, είτε την Πολωνία, το πρόβλημα είναι το ίδιο. Απλώς εδώ έχω αναφέρει τις μεγαλύτερες χώρες με ισχυρέ σχετικά διοικητικές δομές. Το κοινωνικό και το περιφερειακό ταμείο φυσικά εμπλέκονται σε διαφορετικά επιχειρησιακά προγράμματα. Τα κράτη-μέλη προσπαθούν να αντιμετωπίσουν προτεραιότητε, να λάβουν την καλύτερη απόφαση για το ποιο ταμείο ταιριάζει καλύτερα στο ένα ή το άλλο έργο. Τα αποτελέσματα όμω πολλέ φορέ είναι εκπληκτικά. Ε, το ταμείο που υποτίθεται να λαμβάνει ένα συγκεκριμένο ρόλο δεν μπορεί να εμπλακεί στο πρόγραμμα που του ανήκει. Υπάρχει προβλήματα, υπάρχουν προβλήματα συντονισμού, συνέπεια σε παρεμβάσει μια συγκεκριμένη περιοχή. Δηλαδή, μια εθνική αρχή εμπλέκεται με το Περιφερειακό Ταμείο για τη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά η τοπική αυτοδιοίκηση τρέχει ένα πρόγραμμα για το Κοινωνικό Ταμείο στην ίδια περιοχή, χωρί να ξέρει ο ένα ε, τι πει ο άλλο και χωρί να υπάρχει οποιοδήποτε συντονισμό. Ακόμα και μεγάλοι δήμοι πλήττονται από το πρόβλημα από αυτόν τον παραλογισμό. Εν ώψη της Ατζέντα 2020, ε, καλό θα είναι να μισθούν όλα αυτά, ή αλλιώ υπάρχει κίνδυνο να γίνουν όλα αυτά χειρότερα. Ένα άλλο παράδειγμα, εδώ. Παρά την σχετική πολυπλοκότητα, αυτό το περιλάβει εδώ ως παράδειγμα, γιατί στην Αγγλία, έτσι όπως λέει και η Κομισιόν, υπάρχει μια σχετικά, σχετικά καλή κατανομή αρμοδιοτήτων. Παρά το γεγονός αυτό, όμως, βλέπετε εδώ Ακριβώ επειδή υπάρχει η γνωστή διοικητική κατάδυμηση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Βλέπετε στην Αγγλία, για παράδειγμα, έχετε τρία διαφορετικά κανάλια, το Περιφερειακό Ταμείο, με νέα επιχειρησιακά προγράμματα. Μετά έχετε το ενιαίο του κοινωνικού και ένα ξεχωριστό του γεωργικού. Και όλα αυτά τα διαχειρίζονται διαφορετικά υπουργεία. Τώρα, αν είσαστε δήμο που προσπαθείτε να συνδυάσετε όλα τα παραπάνω είναι δεδομένο ότι θα αντιμετωπίσετε προβλήματα ακόμη και αν είστε καλά οργανωμένο ε, δημόσιο και τα έχετε όλα αυτά πολύ καθαρά στο μυαλό σα. Στη Σκωτία και την Ουαλία τα πράγματα είναι λίγο πιο εύκολα λόγω του ότι όλα θα διαχειρίζεται η σκοτική κυβέρνηση που είναι πάλι μια διοίκηση εδώ δεν έχουμε διαφορετικά υπουργεία, αλλά διαφορετικές διευθύνσει αν θέλετε. Ε, είμαστε λίγο πιο, σε πιο οικογενειακό περιβάλλον, αλλά και πάλι διαφορετικοί διευθυντέ, διαχείριζονται τα ίδια πράγματα. Όσο καλέ να είναι η σχέση και η συνεργασία, κάποια πράγματα μπερδεύονται, γιατί πρέπει να τηρούμε τους κανόνες και των δύο ή τριών ταμείων. Αγροτικό τομέα συνοχή. Ίσως πιο δύσκολη περίπτωση. Αν... Γιατί δύο διαφορετικέ γενικέ διευθύνσει εμπλέκονται και πάλι. Έχουμε λοιπόν το Χρονικό Ταμείο, το Ταμείο Εγγύσεων. Πρόκειται για δύο μισοδύναμε σχεδόν ταμεία και ειδικά στον άξονα 3 με το leader ε, διαφορετικά ταμεία, διαφορετικοί μηχανισμοί ασχολούνται με τα ίδια πράγματα. Υπάρχουν βεβαίω και εδώ οι σχετικέ οδηγίε, αλλά ποια είναι η διαχωριστική γραμμή. Αυτή υπάρχει μόνο σε επίπεδο έργου. Άρα δεν αποφεύγονται οι επικαλύψεις, οι γκρίζες ε, ζώνες και εδώ και πάλι για άλλη μια φορά διαφορετικά υπουργεία σε διαφορετικές χώρες ασχολούνται με τα ίδια πράγματα χωρίς πολλές φορές να μιλούν το ένα με το άλλο. Αυτό μας λένε τα μέλη μας. Σε περιφερειακό επίπεδο έχουμε δύο επιτροπές, δύο διαφορετικές επιτροπές παρακολούθησης. Τα μέλη είναι διαφορετικά στην κάθε επιτροπή. Συντονισμό υπάρχει μόνο σε πολύ χαλαρό επίπεδο. Δεν μπορούμε να μιλάμε λοιπόν για ενιαία προσέγγιση. Εδώ ένα κλασικό παράδειγμα είναι όταν το Περιφερειακό Ταμείο και το Αγροτικό Ταμείο εμπλέκονται σε διαφορετικά τμήματα του ίδιου έργου. Εκεί πάλι συγχαίρονται διαχωριστικές γραμμές. Και για να καταλήξω, όπως ίσως ε, Βλέπετε αυτά είναι στα σουηδικά, μην... δεν φτάνει τα αγγλικά σας. Ε, αυτό δίνει μια εικόνα της πολυπλοκότητας που αντιμετωπίζει το τοπικό επίπεδο όταν έχει να δουλέψει με τα εθνικά αλλά και με τα κοινοτικά ταμεία. Εδώ το παράδειγμα αφορά την Σουηδία. Υπάρχει εκεί ένας νόμο ο οποίο επιχρεώνει την τοπική αυτοδιοίκηση να παρέχουν ευρυζωνικές συνδέσεις. Εξετάζουν λοιπόν οι Δήμοι τι λεφτά υπάρχουν εθνικά ή κοινοτικά. Βλέπετε εδώ είναι σαφής η κοινωνικα βλεπετε εδω ειναι σαφης η επικαλυψη των αρμοδιοτήτων μεταξύ ε, όλων των επιπέδων ευρωπαϊκού, εθνικού, περιφερειακού, τοπικού. Υπάρχει επικάλυψη όσον αφορά τον τύπο του προγράμματος. Είναι υποδομές, είναι κοινωνία τη γνώση τι είναι. Άρα λοιπόν και εδώ οι διαχωριστικέ γραμμέ συγχέονται. Βλέπετε για άλλη μια φορά πόσες επικαλύψεις υπάρχουν. Και που να δείτε τι γίνεται με την ε, κοινωνική ένταξη ή την ανάπτυξη τοπικών κοινωνιών κλπ. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Ιδιαίτερα επαναλαμβάνω για έναν μικρό δήμο. Αυτά όλα βεβαίω θα μας πει κάποιος είναι από τη φύση τους ε, πολύπλοκα. Δεν γίνεται αλλιώς. Το θέμα είναι όμως να αντιμετωπίσουμε τοπικά προβλήματα. Χρειαζόμαστε αποτελέσματα. Και μόνο αν όλος αυτός ο μηχανισμός γίνει φιλικός προς τον χρήστη, σε τοπικό επίπεδο μπορούμε να έχουμε κάποια αποτελέσματα. Μόνο έτσι μπορούμε να υλοποιήσουμε πραγματικά ευρωπαϊκά προγράμματα σε τοπικό επίπεδο. Χρειάζεται λοιπόν να διευκολύνουμε του τοπικού πρωταγωνιστές. Επόμενη διαφάνεια. Εν κατακλείδη, Οι ειδικοί συμφωνούν ότι ένα νέο ταμείο θα έκανε τα πράγματα πολύ πιο εύκολα. Γνωρίζουμε από την έκθεση για την συνοχή και την έκθεση για τον προπολογισμό ότι αυτό είναι δύσκολο να γίνει. Το έτοιμα φυσικά παραμένει στο τραπέζι, όμω, για του επόμενου εννέα μήνε έχουμε μια ευκαιρία να καταστρώσουμε ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο. Το συζητούμε με τους ειδικού και η συμβουλή είναι να προσπαθήσουμε το στρατηγικό πλαίσιο να είναι γενικό και να συμπεριλάβει όλα τα ταμεία. Δηλαδή οι επιμέρους κανονισμοί να απλουστευτούν όσο γίνεται ή να συντομευθούν εν πάση περιπτώσει και οι εξαιρέσεις να είναι πράγματι εξαιρέσεις και να μην δίνουν μεγαλύτερο περιθώριο ερμηνεών. Επίσης οι εθνικοί κανόνες πρέπει να γίνουν πιο σαφείς και να μην τροποποιούνται κάθε λίγο και λιγάκι. Εμείς ως ε, CEMR και Κόσλα, βεβαίω, πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνον εφόσον ξεκινήσει κανείς από τη μελέτη των τοπικών προβλημάτων. Και εμεί καλούμε την Κομισιόν μαζί με του ειδικού στο τοπικό επίπεδο να εξετάσουν τα τοπικά προβλήματα μαζί με το CMR και να ε, βρει τρόπους η Κομισιόν να αντιμετωπίσει αυτές τις επικαλύψεις και τις συγχύσεις. Η έκθεση για την συνοχή λέει και αυτή ότι πρέπει να προσφέρουμε ένα νέο υπόδειγμα δράσης για την συνοχή σε τοπικό επίπεδο. Επίσης κάποιοι λένε ότι και το urban πρέπει να ενταχθεί σε αυτό το στρατηγικό σχέδιο. Αλλιώς ε, δεν θα υπάρχει αυτοσυνέπεια. Αν και ξέρω ότι πολλοί θα διαφωνήσουν με αυτό στη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Βέβαια, και αυτό είναι το τελευταίο μου σχόλιο, ο χρόνος πιέζει. Αν μπορέσουμε να ενοποιήσουμε τα ταμεία και να πετύχουμε συνέργειες θα χρειαστεί τεράστια διοικητική δουλειά του επόμενους 9 μήνες. Όταν ε, ασχοληθούμε συγκεκριμένα με το έργο αυτό θα, θα αντιμετωπίσουμε σίγουρα δυσκολίες. Η Κομισιόν πάντως έχει συμβούλους και πάρα πολλές τοπικές ενώσεις περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκηση που μπορούν να βοηθήσουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ήταν ε, πάρα πολύ χρήσιμες ε, οι τρεις απόψεις που ακούσαμε, καθώς είναι και αλληλοσπληρωματικές. Εδώ βρίσκεται ο κύριος Πίτερ Μπέρκοβιτς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο τέλος της συζήτησής μας θα καλέσω και τον κύριο Μπέρκοβιτς ε, να μας εξηγήσει πόσο μακριά μπορούμε να πάμε σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πόσο μακριά σχεδιάζει να πάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με αυτούς τους κοινού ε, κανόνες και τα κοινά συστήματα για όλα τα διαρθρωτικά ταμεία για την ε, επόμενη πολιτική συνοχή. Αλλά τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στους συναδέλφους που το επιθυμούν. Ακόμη δεν έχει ζητήσει κανείς το λόγο. Κύριε Τεξέιρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Σταυρακάκη για το έγγραφο εργασία. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλά δομημένο. Είναι ένα φιλόδοξο και αντικειμενικό έγγραφο όπου το οποίο εστιάζει στα σημαντικά ζητήματα. Εγώ θα ήθελα να τονίσω εδώ πέντε σημεία. Καταρχήν ότι οι συνέργειες μπορούν να έχουν καλά αποτελέσματα σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και μπορούν να έχουν καλύτερα αποτελέσματα από ένα κοινό ταμείο με κοινού κανόνε. Επίση, ε, συμφωνώ ότι αυτό ο συντονισμό πρέπει να γίνει για να υπάρχει συνοχή και συνέργειε. Και στο θέμα τη συνοχή, είναι προφανείς κάποιες πτυχές, κυρίως ό,τι αφορά τη σύνδεση ε, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του ΕΤΠΑ. Εγώ θεωρώ ότι στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ οι οικονομικές πρωτοβουλίες μπορεί να είναι πιο ε, αποτελεσματικές αν συνδεθούν με πρωτοβουλίες για την κοινωνική ανάπτυξη. Επίσης, ε, θα πρέπει να αξιολογήσουμε το θέμα της διαφοροποίησης του Γεωργικού Ταμείου και πρέπει να δούμε αν θα πρέπει να διατηρήσουμε αυτό το διαχωρισμό και αν αυτός ο διαχωρισμός ε, ωφελεί ή όχι για να έχουμε ευκαιρίες ε, ισότιμης ανάπτυξης μεταξύ αστικών περιοχών και περιοχών της υπαίθρου. Κατόπιν ε, αυτή η ανάγκη μεγαλύτερου συντονισμού είναι κάτι αναπόφευκτο σήμερα. Αυτό λόγω της οικονομικής κρίσης που ζητεί αυτή τη στιγμή η Ευρώπη και αυτό μας οδηγεί στο αναπόφευκτο, στην αναπόφευκτη λύση. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα με τα διαθέσιμα μέσα. Και αυτή είναι ε, η κατάλληλη χρονική στιγμή για να το πράξουμε, όχι αργότερα. Και πέμπτον, συμφωνώ ότι αυτός ο συντονισμός πρέπει να γίνει σε όλα τα επίπεδα και με ένα οριζόντιο και ε, εγκάρσιο τρόπο. Πρέπει να συμμετέχουν όλες οι αρχές και οι τοπικές αρχές και πρέπει να έχουμε συμμετοχή όλων των επιπέδων και εν τέλει να έχουμε και έλεγχο και αξιολόγηση. Αυτό μου με οδηγεί στο να υπενθυμίσω ότι η συνθήκη δεν ε, προβλέπει μόνο αυτή την κοινή δράση για τα διαφορετικά ταμεία, αλλά και άλλα διαθέσιμα μέσα. Θέλω εδώ να υπενθυμίσω το ρόλο τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το κάνω αυτό για έναν απλό λόγο, γιατί εδώ έχω μία είδηση από μια υποδομή που θα αναπτυχθεί ε, στο ε, Μαρόκο, στην ε, Ταγκερή. Θα έχουμε μια επένδυση 200 εκατομμυρίων για να γίνει το λιμάνι της σε ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Μεσογείου. Και αυτό είναι ενισχυτικό, αν μου επιτρέπετε, γιατί είναι σχεδόν σχιζοφρενικό σε μια χρονική συγκυρία όπου έχουμε ανεργία σε όλη την Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, θα επενδύσει τόσα χρήματα σε ένα λιμάνι που τελικά θα καταστήσει μη ανταγωνιστικά τα λιμάνια Πορτογαλίας, Ισπανίας και Ιταλίας και ξέρουμε ότι σε αυτό το λιμάνι έχει αναπτυχθεί αθέμητος ανταγωνισμός γιατί ε, λειτουργεί με κοινωνικό ντάμπινγκ και μάλιστα σε μια συγκυρία όπου πρέπει να λάβουμε μέτρα για την καταπολέμηση της ενεργείας βλέπουμε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να χρηματοδοτεί τον κύριο ανταγωνιστή των Ευρωπαϊκών Λιμανιών. Και έτσι λοιπόν αυτό το θέμα της, του συντονισμού και των συνεργειών δεν μπορεί να είναι κάτι θεωρητικό. Εδώ τι μετράει, δεν μετρά ε, μόνο ε, η θεωρητική οικοδόμηση, αλλά πρέπει να υπάρχει και δέσμευση και υλοποίηση. Δηλαδή, πέρα από το να συζητούμε τώρα εμεί θεωρητικά εδώ με ποιο τρόπο μπορούμε να έχουμε συντονισμό και συνέργειε, αυτό που πρέπει να κάνουμε στην πραγματικότητα είναι να εφαρμόσουμε και να εκτελέσουμε αυτό το συντονισμό και τι συνέργειε. Ευχαριστώ. Yes. Now it's here. Yeah. Thank you very much for... Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Σταυρακάκη για την έκθεση αυτή. Πιστεύω ότι είναι πολύ σοβαρό το θέμα και πρέπει να συζητηθεί. Από ό,τι κατάλαβα, η κύρια πρόταση που συνιστά μια καθολική πρόταση είναι στη σελίδα 6 όπου μπορούμε να δούμε ότι θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλίας και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο να ενταχθούν στην ίδια δομή που είχαμε στην περίοδο 2000-2006. Εγώ νομίζω ότι αυτή είναι πάρα πολύ σοβαρή πρόταση και η, ερώτησή μου ε, απευθύνεται ίσως σε κάποιον από την Κομισιόν. Αν δούμε ε, τρόπο υπολογισμό το δεύτερο πυλώνα του Γεωργικού Ταμείου η ανάπτυξη, η αγροτική ανάπτυξη δεν έχει χρησιμοποιηθεί καταλήλω τα τελευταία 3-4 χρόνια. Το 2009 80% των χρημάτων, δηλαδή 1,8 δισεκατομμύρια, δεν πληρώθηκαν και ε, ουσιαστικά δόθηκαν σε σχέδια οικονομικής ανάπτυξης. Τώρα σε αυτόν τον τροποποιητικό προπολογισμό η Επιτροπή Προπολογισμού σχετίζει να πάρει ένα δισεκατομμύριο από το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και να τα χορηγήσει στα διευθυντικά ταμεία, δηλαδή στο Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και στο Ταμείο Συνοχής. Η ερώτηση λοιπόν είναι πρόκειται να συγχωνεύσουμε αυτό το σύστημα διαχείρισης για να πάρουμε μόνο ένα τμήμα και μιλώ για το δεύτερο πυλώνα, αγροτική ανάπτυξη και έχουμε περίπου 12 δισεκατομμύρια το χρόνο εκεί. Εγώ ε, ε, στην πατρίδα μου τέθηκε συζήτηση οι άνθρωποι γιατί δεν ε, αντιδρούν ε, ε, η απάντηση είναι ότι οι αγρότες χρειάζεται χρήματα για τη χρηματοδότηση. Δεν δίνονται αυτά τα χρήματα από το κράτος, δεν έχουν ε, και χρήματα από τις τράπεζες, αλλά δεν ενδιαφέρονται. Ενδιαφέρονται για τον πρώτο πυλώνα, για τις πληρωμές ανεκτάριου, για τις άμεσες πληρωμές. Αλλά η ερώτηση είναι, εδώ σχεδιάζουμε πληρωμές 12 δισεκατομμυρίων το χρόνο που δεν δαπανώνται σωστά και η ερώτησή μου είναι και στον εισηγητή, ίσως είναι πιο ρεαλιστικό να μιλήσουμε για συνέργειες. Αν πάρουμε το δεύτερο πυλώνα, γιατί νομίζω δεν είναι ρεαλιστικό να μιλάμε για τον πρώτο πυλώνα, γιατί σχετίζεται με τις πληρωμές ένα εκτάριο περισσότερο και όχι, περισσότερο, και όχι τόσο με την ανάπτυξη συνολικά. και ίσως κάτι ακόμα, ότι έχουμε διαφορετικές καταστάσεις ε, ή αγροτικές συμφωνίες σχεδόν και 10 χρόνια, δηλαδή κατά μία 7 έτη. Αν μιλούμε τώρα ε, για το μέλλον του MFF, τότε πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τις δημοσιονομικές προοπτικές. Υπάρχουν ε, λοιπόν διαφορές σε ό,τι αφορά την οριμότητα. Έτσι λοιπόν υποστηρίζω την πρόταση του συγητή, όμως ίσως να μην μιλάμε για το σύνολο του το Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου, αλλά για ένα πυλώνα όταν μιλάμε για την αγροτική ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. πολύ ενδιαφέρον η όλη παρουσίαση και φυσικά η εισήγηση και όλα αυτά που ακούσαμε πριν και εμπλουτίζουν πραγματικά τη λειτουργία της ε, Επιτροπής θα ήθελα να επισημάνω και εγώ κάποια σημεία από το έγγραφο εργασίας του εκλεκτού συναδέλφου του κ. Σταυρακάκη. Πραγματικά ε, η τρέχουσα κατάσταση, οι προοπτικές αλλά και οι μελλοντικές ε, συνέργειες για αυξημένη αποτελεσματικότητα μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και άλλων διαρθρωτικών ταμείων είναι έννοιες που οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιμένουν να δουν στην πράξη και είναι πολύ κρίσιμη ε, αυτή η συζήτηση χρονικά εν μέσω δηλαδή μιας ε, κρίσης που περνά η Ευρωπαϊκή Ένωση και με τα γνωστά και συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλές περιφέρειες. Βέβαια, σαφώς και πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι, να μην ε, κινούμαστε σε αοριστείες. Οι μέχρι τώρα επιδόσεις ε, θα μπορούσα να πω ότι είναι ελαφρώς ικανοποιητικές αλλά θέλοντας να παραμείνω αισιόδοξο, θα νιώθω ότι πρέπει να τονίσω ότι δεν πρέπει να εφησυχάζουμε ε, να ανεβεί, πρέπει να ανεβεί η ταχύτητα θα πρέπει ε, να συμφωνήσω νιώθω ότι πρέπει να συμφωνήσω με τον συντάκτη στα εξή σημεία η χρηματοδότηση των οικονομικών δραστηριοτήτων πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν με επίκεντρο τον άνθρωπο τις τοπικές οικονομίες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή ακόμα και τις ιδιαιτερότητές τους. Πράγματι, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας και των δύο διαρθρωτικών ταμείων συνδέεται με την πρόοδος προς την επίτευξη συνέργειας μεταξύ οικονομικής και κοινωνικής παρέμβασης. Οι νέοι κανόνες διασταυρούμενης χρηματοδότησης πρέπει να αναθεωρηθούν ουσιαστικά. Και φυσικά αφού ε, βγουν πρώτα τα ε, χρήσιμα συμπεράσματα που χρειάζεται. Προφανώς και πρέπει να πει κανεί ναι στις συνέργειες, αλλά επιμένω και πάλι πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι. Και υπάρχει το ερώτημα, θέλουμε απλά τη συμμετοχή και συνέργεια των ταμείων στοχευμένη σε μια συγκεκριμένη πολιτική και ένα πρόβλημα που μας απασχολεί ή επιθυμούμε συμμετοχή και συντονισμό σε ένα ευρύτερο αναπτυξιακό πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει διάφορους τομείς πολιτικής. Φυσικά υποστηρίζω την, ε, το δεύτερο δρόμο όπου έτσι πολύπλευρα προβλήματα θα βρουν αποτελεσματικότερη λύση με βιώσιμο και με μακροπρόθεσμο τρόπο. Άλλωστε, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε εστιάσει επανειλημμένα, όπως βλέπουμε και στην πέμπτη έκθεση της Επιτροπής για τη Συνοχή, ότι στοχεύουμε πάντα σε μια ενιαία, ευέλικτη πολιτική σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κλείνοντας λοιπόν, χαιρετίζω το έγγραφο εργασίας και όλη την ενδιαφέρουσα διαδικασία και περιμένω με ενδιαφέρον και από, τους, ε, από το σώμα ε, και με βάση τις εμπειρίες που πρέπει να εμβαθύνουμε και να δούμε στην πράξη την αποτελεσματικότητα αυτών των πολιτικών. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να σχολιάσει τη συζήτησή μας, τον κύριο Σπικοβίτς. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον εισηγητή για τον έγγραφο αυτό, το οποίο είναι συνοπτικό αλλά πάρα πολύ πλούσιο ε, και εκφράζονται πολύ ενδιαφέρουσες ε, ιδέες. Θέλω να είμαι σύντομο. Υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικά σημεία που τέθηκαν από τους ε, ομιλητές, αλλά θέλω να τονίσω τα κύρια στοιχεία του σκεπτικού της Κομισιόν, κυρίως στο πλαίσιο του εγγράφου της αναθεώρησης του προπολογισμού και της πέμπτης έκθεσης συνοχής. Νομίζω ότι η Κομισιόν προωθεί ιδέες για τη βελτίωση της ολοκλήρωσης και των συνεργειών σε τρία επίπεδα. Καταρχήν στο πλαίσιο ενός κοινού στρατηγικού πλαισίου για τις επενδύσεις που θα καλύπτει πέντε ταμεία δηλαδή το Κοινωνικό Ταμείο, την Αλία, ε, το βιτρονικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης λοιπά, Αλλά θα υπάρχει σύνδεση και θα μπορούσε να υπάρχει σύνδεση με άλλα μέσα. Σε εθνικό επίπεδο θα υπάρχουν ε, μάλλον θα προτείνονται συμβάσεις εταιρικής σχέσης και αυτό σημαίνει δηλαδή συμφωνία μεταξύ ευρωπαϊκού επίπεδου και των φορέων που θα είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για την επίτευξη των στόχων. Η κάλυψη αυτών των συμβάσεων προτείνεται να είναι για την πολιτική συνοχή, αλλά επίσης είναι ανοιχτό και το ζήτημα αν θα επεκταθεί και σε άλλα ταμεία. Και τέλος, στην έκθεση της συνοχής τονίζεται ότι αυτές οι συμβάσεις εταιρικής σχέσης θα περιγράφουν και τους μηχανισμούς συντονισμού μεταξύ των ταμείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε το επίπεδο, σε επίπεδο δικαιούχων. Η Κομισιόν είναι ιδιαίτερα ανήσυχη για ε, πιθανές πολυπλοκότητες που μπορούν να προκύψουν σε ό,τι αφορά τους κανόνες επιλεξιμότητας και στο έγγραφο αναθεώρηση του προπολογισμού προτείνεται μία εναρμόνιση κανόνων επιλεξιμότητας και εφαρμογής και για τους κοινούς κανόνες όπου είναι δυνατό μεταξύ των διαφορών χρηματοδοτικών μηχανισμών και αυτό το εγχείρημα έχουμε αναλάβει τώρα με την Κομισιόν κατά την εκπόνηση των ε, νομοθετικών μας προτάσεων. Θέλω να τονίσω δύο σημεία που εξετάζουμε αυτή τη στιγμή που έχουν να κάνουν και με κάποια σημεία που ανεφεραν οι ομιλητές. Καταρχήν την ιδέα ότι θα πρέπει να έχουμε μία ε, και μόνο προσέγγιση για την τοπική ανάπτυξη και στα τέσσερα ταμεία που ε, προωθούν τώρα την τοπική ανάπτυξη, δηλαδή και στο Ταμείο Αλίας ε, και Αγροτικής Ανάπτυξης και στο Κοινωνικό Ταμείο και στο ΕΤΠΑ θα έπρεπε οι δικαιούχοι να έχουν μία και μόνη προσέγγιση για να αποφεύγεται ο πολλαπλασιασμό των κανόνων. Ένα δεύτερο θέμα που τονίστηκε είναι το θέμα της διασταυρούμενης χρηματοδότησης. Η διασταυρούμενη χρηματοδότηση είναι σημαντικό ζήτημα γιατί επιτρέπει στους δικαιούχους σε τοπικό επίπεδο να επιλέξουν τον καλύτερο τρόπο συνδυασμού των ε, κονδυλίων ε, για την ε, επίτευξη των στόχων. Ε, οι σημερινοί κανόνες διασταυρούμενη χρηματοδότηση είναι ίσως υπερβολικά πολύπλοκοι και θα μπορούσαν να βελτιωθούν ή να απλουστευτούν. Αυτός λοιπόν είναι ένα τομέα που εξετάζουμε. Και θέλω και να τονίσω το πόσο σημαντικό θεωρούμε την κοινή χρηματοδότηση πρωτοβουλειών, κυρίως σε τοπικό επίπεδο. Ίσως ε, το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό πλαίσιο είναι η πλατφόρμα κατά της φτώχειας. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό εκεί να συγκεντρώσουμε τα διάφορα ταμεία έτσι ώστε να εργαστούμε με ένα ολοκληρωμένο τρόπο και στην Ήπεθρο αλλά και στα αστικά κέντρα. Και τέλος, έχουμε επιτάπητος και μία πρόταση αναθεώρησης του χρηματοδοτικού μηχανισμού κανονισμού, με συγχωρείτε. Το θέμα που τέθηκε είναι η εναρμόνιση των ελέγχων και η αναθεώρηση του χρηματοοικονομικού κανονισμού προτείνει εν μέρη εναρμόνιση των ε, μηχανισμών ε, εγγύσεων για τις ε, πολιτικές κοινή διαχείρισης. Όμως εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες για την εναρμόνιση, γιατί στη συζήτηση πολλοί από ε, τους ενδιαφερομένους τόνισαν τις διαφορές που υπάρχουν ε, μεταξύ ε, των δαπανών ε, διαρθρωτικών ταμείων και των αγροτικών δαπανών. Αυτά υπάρχουν επιτάπητος για να συνοψίσω τρία στοιχεία ε, σκέφτεται η Κομισιόν μια πιο στρατηγική προσέγγιση για το να θέσει προτεραιότητες ε, στα ταμεία, να απλουστεύσει τη διαχείριση των ταμείων μέσω της εθνικής διοίκησης, να διευκολύνει την πρόσβαση στα ταμεία, την πρόσβαση των δικαιούχων στα ταμεία ε, σε επίπεδο επιχειρησιακό. Πολλά θα μπορούσαμε να κάνουμε σε επίπεδο ευρωπαϊκού κανονισμού, αλλά εγώ νομίζω ότι και τα κράτη-μέλη και η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να διαδραματίσουν το δικό τους ρόλο. Ακούστηκα κάτι σε σχέση με το κατακαιρματισμό των δομών ε, σε εθνικό επίπεδο. Αυτό είναι ένα θέμα που αφορά τα κράτη-μέλη, είναι ένα θέμα επικουρικότητας και Επίσης είναι σημαντικό οι αρμόδιοι φορείς για την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής ε, να χρησιμοποιήσουν πλήρω τις ευκαιρίες ε, για να καταλήξουν στα επιθυμητά αποτελέσματα. Ευχαριστώ Πίτερ. Γιώργο θες να πεις δύο λόγια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους ε, προσκεκλημένους ομιλητές για τις πολύ ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις τους και παρουσιάσεις τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης θερμά τους συναδέλφου για τις πρώτες θετικέ. Ε, παρατηρήσεις και σχόλιά τους. Ευελπιστώ ότι όλοι οι συνάδελφοι θα συμβάλλουν επικοδομητικά με τις απόψεις τους, τις προτάσεις τους, τα σχόλιά τους, τη διαμόρφωση της έκθεσης. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την έκθεση. Σχεδιάζουμε ε, να εγκριθεί το Φλεβάρι. Να πω ότι για άλλη μια φορά ότι εκτιμούμε ιδιαίτερα τη συμβολή των προσκεκλημένων μας ε, γιατί μας βοήθησαν να κατανοήσουμε καλύτερα την πλευρά των ανθρώπων που εφαρμόζουν στην πράξη ε, αυτά τα προγράμματα και αυτό διευκολύνει και την αύξηση της αποτελεσματικότητας της χρήσης των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Ο Πίτερ Μπέρκοβιτς επίσης ανέφερε την ισχυρή δέσμευση της Κομισιόν να προχωρήσουν περαιτέρω σε αυτό τον δρόμο της καλύτερης αποτελεσματικότητας των πολιτικών και καλύτερη, της καλύτερης ευθυγράμμισης και εναρμόνισης που θα επιτρέψει τις συνέργειες μεταξύ των διαφόρων μορφών χρηματοδότησης. Ελπίζω ότι θα μείνετε πιστεί και θα παρακολουθήσετε την συζήτηση που θα γίνει στην Επιτροπή μας και στο Κοινοβούλιο για αυτό το θέμα για τη δομή της μεταλλοντικής πολιτικής η οποία θα διαρθωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μας επιτρέψει να χρησιμοποιήσουμε τις επενδύσεις που έρχονται από τα διαρθρωτικά, κονδύλια. Και τώρα έχουμε μια δημόσια ακρόαση για τη θέση των ευρωπαϊκών πόλων και αστικών κέντρων στην πολιτική της συνοχής. Ο χρόνος μας είναι μέχρι τις 11.45 για αυτή τη συζήτηση. Έχουμε πέντε ομιλητές, δύο συναδέλφους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ξεκινήσουμε με αυτούς. Επίσης έχουμε τις Eurocities και το έναν εμπειρογνώμονα από το Πανεπιστήμιο της Πράγας, ε, ο οποίος είναι εδώ μαζί μας, όπως επίσης ε, και από ένα ερευνητικό ίδρυμα από τη Βουδαπέστη υπάρχει εμπειρογνώμονας. Ε, δεν έχουμε τον Μπισέλ ΠΑΚ σήμερα εδώ και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση να ξεκινήσουμε με τον Ντάνιελ Μουκέ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο οποίο θα μιλήσει για το παρελθόν, για την αξιολόγηση του, της κοινοτικής πρωτοβουλίας Urban 2000-2006. Έχουμε πολύ χρόνο, αλλά όχι όσο θα θέλαμε, οπότε ας είστε όσο πιο σύντομοι γίνεται. Πείτε μας μόνο τα σημαντικά. Ντανιέλ Μουκέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχω μία παρουσίαση, έρχεται στις οθόνες σας. Ευχαριστώ να ξεκινήσω ε, κάνοντας μια εισαγωγή στην κοινωνική πρωτοβουλία για το Urban 2. Ε, πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Τι ήταν το Urban 2, για όσους ε, δεν το γνωρίζετε, ήταν ένα εργαλείο που μας βοήθησε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα των αστικών ε, γειτονιών σε κρίση. Τι εννοούμε γειτονιά σε κρίση, μια περιοχή με μεγάλη ενεργεία, με ένα φυσικό περιβάλλον που βρίσκεται σε παρακμή, ε, κάποιο έλλειψη πρασίνου και κοινωνικά προβλήματα, ο έγκλημα κτλ. Όλα αυτά συνδυάζονται σε μια ε, αστική περιοχή. Υπήρξαν 17 ε, προγράμματα στα παλιά κρατημέλη. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό μας είναι ότι πρόκειται για σχετικά μικρές περιοχές. Κοιτάξτε αυτό τον αριθμό των, προγραμμα... των ανθρώπων διαιρεμένο δια 70 έχουμε, ε, δια 17 ε, συγγνώμη, έχουμε ε, σχεδόν 3.000 άτομα. Έχουμε λοιπόν σχετικά μικρές περιοχές ε, που τα προβλήματα είναι συγκεντρωμένα. Αν δείτε λοιπόν τη χρηματοδότηση και κάνετε τα μαθηματικά θα δείτε ότι η ένταση των ενισχύσεων ήταν σχετικά μεγάλη. Κατά μέσο όρο ήταν παρόμοια με αυτήν του στόχου 1 στην ίδια περίοδο. Μικρές περιοχές, ε, μεγάλη ένταση προβλημάτων, μεγάλη ένταση ενισχύσεων η μέθοδος Urban ήταν η παροχή μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης ε, για την αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων οικονομικών, κοινωνικών ε, και προβλημάτων ε, παρακμής του φυσικού περιβάλλοντος. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν οι ισχυρέ εταιρικέ σχέσεις σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή σχέσεις με την τοπική κοινότητα, το Δήμο, γενικά όλους τους φορείς ε, που σχετίζονται ε, με τις δράσεις σε τοπικό επίπεδο. Επόμενη διαφάνεια. Κάποιες βασικές στατιστικές. Αν ε, κρατήσετε στο μυαλό σας μία λέξη που έχει σημασία είναι ότι η αξιολόγηση ήταν εις βάθος. Μία αξιολόγηση εις βάθος και των 17 προγραμμάτων, αν δείτε την τεκμηρίωση, τα δεδομένα, τις στατιστικές και τα δεδομένα προγράμματος, Υπάρχουν πάρα πολλά διαθέσιμα, υπάρχουν 15 μελέτες περίπτωσης που επιλέξαμε και φτιάξαμε ένα ισορροπημένο δείγμα για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο εκπροσωπεί ένα αγμίγμα ισορροπημένο των διαφόρων στρατηγικών και προσεγγίσεων, όπως και μείγματα σε άλλα επίπεδα, κάποια σε μεγάλες πόλεις, κάποια σε μεσαίας κλίμακας και μικρές πόλεις. Με άλλα λόγια, αυτές οι 15 μελέτες περίπτωσης ήταν όσο αντιπροσωπευτικές γινότανε οι μελέτες εις βάθος αυτές ε, είχαν να κάνουν με μια ε, επίσκεψη τριών εβδομάδων που ε, ερχόμασταν σε επαφή με τους τοπικούς φορείς και κοιτούσαμε τι ακριβώς γινόταν, φτιάχναμε και μικρές μελέτες περίπτωσης και τα αποτελέσματα φιλτράρονταν από τρεις επιστημονικούς εμπειρογνώμονες και φτιάξαμε ένα ε, ισορροπημένο πάνελ, το Michael Πάρκινσον ο οποίος είναι υπέρ του Urban, αλλά και κάποιους που ήταν σκεπτικιστές, έναν Ιταλό καθηγητή ας πούμε, ο οποίος ήταν στο άλλο άκρο και κάποιον ενδιάμεσα. Είχαμε λοιπόν αυτούς τους τρεις διαφορετικού ε, εμπειρογνώμονε που έκαναν την έκθεσή τους και θέσαν υπό τα αποτελέσματα και τα ενέκριναν. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια να σας δείξω τα βασικά στοιχεία των χρηματοδοτήσεων. Τα έχω χωρίσει στην ε, φυσική αναγέννηση, την ε, ανοικοδόμηση της οικονομίας ε, και την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού. Πράγματα που δεν είναι εύκολο να διαχωρίσουμε ούτε σε επίπεδο προγράμματος ούτε σε επίπεδο σχεδίου project. Να σας δείξω ε, κάποια βασικά παραδείγματα. Ε, ένα από τα project που εγώ ας πούμε επισκέφτηκα ήταν ένα κτίριο το οποίο ήταν υποδιάλυση. Έγινε κάποια χρησιμοποιήθηκαν ε, τα χρήματα για να χρησιμοποιηθεί το κτίριο αυτό για αυτούς που ήταν μακροχρόνια άνεργοι και ανακαινίστηκε το κτίριο. Και όλα αυτά ήταν μια φυσική, οικονομική και κοινωνική αναγέννηση ταυτόχρονα. Παρ' όλα αυτά, για την παρουσίασή μου θα τα χωρίσω αυτά τα τρία. Πάμε στη φυσική αναγέννηση. Υπάρχουν πολλοί αριθμοί εδώ. Δεν θα σας αφήσω πολύ. Θα σας πω είναι τα 2,3 εκατομμύρια ε, κυβικά, ε, ε, τετραγωνικά ανανεωμένων και ανακαινισμένων κτηρίων. Υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή στο τοπικό περιβάλλον. Αν πάτε σε μια περιοχή urban τώρα θα δείτε κτίρια ανακαινισμένα, χώρους πρασίνου που δημιουργήθηκαν, πάρκα και πεζοδρόμους. Οι περιοχές είναι ξεκάθαρα διαφορετικές από ό,τι ήταν πριν την έναρξη του προγράμματος. Πάμε τώρα στην οικονομική αναγέννηση. Η ανοικοδόμηση της τοπικής οικονομίας και πάλι πολλά τα νούμερα. Ε, όμως ε, υπάρχουν μικρομέτρα τα οποία βοήθησαν τις μικρές επιχειρήσεις ε, τα μαγαζιά, το, να δώσουν επιχειρηματικές υπηρεσίες, να φτιάξουν φυτόρια σε μακροοικονομικό επίπεδο μικροοικονομικό επίπεδο. Ε, μικροοικονομικό γιατί ουσιαστικά εξετάζουμε τις στατιστικές ε, για την περιοχή αυτή και αυτό που είδαμε ε, και μας εξέπληξε είναι ότι τα επίπεδα ανεργίας και στατιστικές ουσιαστικά ακολουθούσαν την οικονομία της ε, πόλης στην οποία βρισκόμασταν. Αν ήταν καλή οικονομία, η ανεργία ας πούμε, στην πόλη ήταν και στην συγκεκριμένη περιοχή. Αυτό λοιπόν δείχνει την τα όρια της τοπικής ε, ανάπτυξης. Μπορεί να αλλάζουμε τη μικροοικονομία, της μικρές επιχειρήσεις, αλλά αν θέλουμε να αλλάξουμε την οικονομία μιας ε, περιοχής, πρέπει να αλλάξουμε την ε, πόλη μέσα στην οποία περιλαμβάνονται. Να πάμε δηλαδή σε ένα πολύ μεγαλύτερο επίπεδο. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια, τη μετώπιση κοινωνικού αποκλεισμού. Και εδώ πάλι έχουμε κάτι που είναι σχεδόν ξεκάθαρο και απτό αν περπατήσετε σε μια περιοχή urban και ρωτήσετε τον κόσμο θα ανακαλύψετε ότι αυτόματα μιλάν για την περιοχή Urban 2 υπάρχουν στοιχεία λοιπόν που δείχνουν την κατάρθιση, τα νέες κοινωνικές υπηρεσίες που προσφέρθηκαν. Σε μια μικρή περιοχή είναι δυνατό με τόσο λίγα χρήματα να αλλάξουμε το έγκλημα και τα ποσοστά ε, του εγκλήματος, να φτιάξουμε καλύτερο φωτισμό στους δρόμους κτλ. Αυτές είναι οι επιπτώσεις λοιπόν σε επίπεδο οικονομίας, φυσικής αναγέννησης και κοινωνικού αποκλεισμού. Να περάσω τώρα σε κάποια από τα οριζόντια συμπεράσματά μας. Αυτό ίσως είναι το κύριο έβριμα, το έβριμα κλειδί της αξιολόγησης, ότι η επιτυχία των project ε, ήταν, ε, ήρθε μέσα από τους ε, τοπικούς από τους κατοίκους σε τοπικό επίπεδο, αυτοί που έλαβαν μέρος ε, και στην εφαρμογή αλλά και στην αποδόση των προγραμμάτων. Και αυτό είναι ένα έβριμα ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Για μένα ως οικονομολόγο, ε, ε, μάλλον ένα συγκεκριμένο προφίλ project θα ήταν αυτό που θα είχε επιτυχία. Δηλαδή, τελικά όμως αυτό που μετράει δεν είναι το τι κάνεις, αλλά το πώς το κάνεις να το κάνεις με τον τόπιο πληθυσμό. 80% των project ε, έτρεξαν από, την από τις τοπικές αρχές και αυτό χαρακτήριζε και το 80% των εταιρικών σχέσεων οι οποίες ε, περιελάμβαναν μια μεγάλη σειρά τοπικών ε, φορέων και αρχών. Η τοπική εταιρική σχέση ναι, μεν έχει σημασία, αλλά τι γίνεται με του μεγάλου παίκτε. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Υπάρχει ένα κρίσιμο ρόλο που μπορούν να παίξουν και αυτοί. Αυτοί δίνουν τι γνώσει και την ικανότητα που χρειάζεται για την εφαρμογή. Οι ντόπιοι έχουν γνώσει σε τοπικό επίπεδο, αλλά δεν ξέρω αν έχουν την κατάρτιση, την δυνατότητα να τρέξουν τα προγράμματα μόνοι τους. Χρειάζονται τέτοια εκπαίδευση. Ένα από τα βασικά στοιχεία που ανακαλύψαμε είναι ότι ενισχύθηκε αυτή η δυνατότητα των τοπικών παικτών να τρέξουν τα προγράμματα. Και αυτό δείχνει και την ε, βελτίωση και τη βιωσιμότητα των project. 60% των project Urban 2 συνεχίζουν μετά από την ε, λήξη του προγράμματος ε, Urban 2. Και αυτό είναι πραγματικά ε, εκπληκτικό, γιατί ούτως ή άλλως ε, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν πρέπει να συνεχίσουν και μετά το τέλο του προγράμματο, όπω η ανακαίνιση ε, ενό κτίριου, για παράδειγμα, αλλά ε, όταν έχουμε ένα ποσοστό 60% τελικά ανακαλύπτουμε ότι είναι εκπληκτικά τα αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν η ανακαινιση ενο κτιριου για παραδειγμα αλλα οταν εχουμε ενα ποσοστο 60 τελικα ανακαλυπτουμε οτι ειναι εκπληκτικα τα αποτελεσματα ετσι λοιπον η πρωτοβουλια των ντόπιων οι οποίοι ενεπλάκησαν ε, στην εφαρμογή ε, είναι αυτοί που χαρακτήρισαν το επιτυχημένο πρόγραμμα, ε, το επιτυχημένο σχέδιο, αλλά ήταν και ένας μεγάλος παίκτη ο οποίος έβαλε την υπογραφή του. Η τελευταία σχεδόν διαφάνειά μου. Να πω ότι ως αξιολογητής δεν θα έκανα το καθήκον μου αν δεν σας πιστούσα την προσοχή σε ένα έβριμα που δεν αφορά μόνο στα Urban 2 αλλά σε πολλά προγράμματα έχουμε προβλήματα με την παρακολούθηση των project, την ιχνηλάτησή τους. Ξεκινάν πάντοτε φιλόδοξα. Ε, υπήρξε ένα σχεδιασμός για 4.000 δείκτες αρχικά. Για μένα αυτό είναι μάλλον ε, υπερβολικό θα έλεγα. έχουμε 59 ε, δείκτες ανά πρόγραμμα, τι γίνεται φυσικά. Το 1 τρίτο αυτών ποτέ δεν καλύπτονται γιατί ξεκινάμε φιλόδοξα, ε, μετράμε, αλλά στο τέλος δεν μετράμε όσα θέλουμε. Η λογική παρέμβαση πολλές φορές επίσης δεν ήταν ξεκάθαρη, ήταν προβληματική σε κάποιες περιπτώσεις. Ένας από τους μάνατζερ του προγράμματος, όταν τον ρώτησαν ποιο είναι το πρόβλημα της περιοχής, είπε ότι ήταν η μακροχρόνια άνεργη. Τι, έκανε, ανακαίνισε το κέντρο της πόλης. Πώς επηρέασε αυτό του μακροχρόνια άνεργους, δεν έχω καμία ιδέα. Δεν μπορώ να σας πω. Έτσι λοιπόν πολλές φορές υπάρχουν οι ανάγκες, έχουν τα χρήματα, αλλά το πρόγραμμα τελικά δεν εστιάζει τις ανάγκες. Και δεν υπάρχει και τρόπος να εντοπίσουμε την πρόοδο. Και αυτό δεν αφορά μόνο στο Urban 2, αλλά και σε πολλά διαφορετικά προγράμματα των διορθωτικών ταμείων. Είναι πολύ σημαντικό να μπορεί κανείς να παρακολουθεί την πρόοδο, να γνωρίζει ποιε είναι οι ανάγκες και να ξέρει τι κάνει και πώς θα αντιμετωπίσει τις ανάγκες, για να μπορέσει κανείς να βρει εάν υπάρχει πρόοδο και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκε. Έτσι λοιπόν ένα από τα συμπεράσματα και τις συστάσεις που θα έκανα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ξεκάθαρη λογική παρέμβαση στα προγράμματα αυτά με κάποιους ελάχιστους καλά επιλεγμένους δείκτες και καλή χνηλάτιση. Αλλά αυτό ίσως είναι ο ρόλος των μεγαλύτερων παικτών. Αυτοί θα βοηθήσουν τους ντόπιου να το κάνουν. Και εδώ έρχομαι στην τελική μου καταληκτική διαφάνεια. Σύμφωνα με στην οποία μπορώ να σας πω ότι αν κοιτάξουμε τις περιοχές Urban 2 υπάρχει μια ξεκάθαρη βελτίωση στην περίοδο 2000-2006. Τα βλέπουμε στις ε, βασικές στατιστικές αλλά και στις μελέτες περίπτωσης. 13,5 από τις 15 μελέτες περίπτωσης ξεκάθαρα υπήρχε πρόοδος. Το Somerville ήταν το πρόβλημα, ήταν καλό το πρόγραμμα, αλλά η τοπική οικονομία ε, κατέρευσε αυτή την περίοδο και πάλι εδώ δείχνεται πώς η, καταδεικνύεται πώς η ευρύτερη οικονομία επηρεάζει τις μικρότερες περιοχές. Υπάρχουν παρόλα αυτά, ε, υπάρχει η βελτίωση, αλλά υπάρχει και όριο σε αυτή τη βελτίωση. Ε, εν μέρει επειδή καλύπτονται μικρές περιοχές, δεν μπορούν να γίνουν όλα. Οι ντόπιοι δεν γνωρίζουν πολλά εκτός της περιοχής τους και απαραίτητα δεν μπορούμε να, να ε, επηρεάσουμε την ευρύτερη οικονομία από μια μικρή περιοχή. Μπορούμε παρόλα αυτά να κάνουμε πολλά, ξεκινώντας από μια μικρή περιοχή, αν συμπεριλάβουμε τους ντόπιου, ε, τους κατοίκους, τους παίκτες ε, και αυτούς που εργάζονται για την κοινότητα και αν έχουμε εμπειρογνώμονες οι οποίοι θα βοηθήσουν τους ντόπιου να δημιουργήσουν τις γνώσεις και τις ικανότητες που χρειάζονται για να τρέξουν τα προγράμματα. Τέλος, ξεκάθαρο είναι ότι πρέπει να γνωρίζουμε τι θέλουμε να κάνουμε, πώς θα είναι η επιτυχία, πώς θα, είναι όταν θεωρηθεί, πώς θα θεωρείται επιτυχημένο και πώς θα το κάνουμε. Ευχαριστούμε πολύ, Ντανέλη και... Θα είμαι λίγο απότομη. Προσέξτε το χρόνο αν θέλετε να έχουμε συζήτηση με τους βουλευτές. Παρακαλώ λοιπόν όλοι, 10 το πολύ για να έχουμε χρόνο για συζήτηση. Ο κ. Νάου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επικεφαλής Μονάδας του Urban. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα με την παρουσίασή μου. Καταρχήν, να υπενθυμίσω γιατί ενδιαφέρομαστε για τις πόλεις. Δεύτερον, να σας πω για την εμπειρία μας από το Urban κατά τη διάρκεια της ε, τρέχουσας προγραμματικής περίοδου και δύο λόγια στην επόμενη διαφάνεια θα συζητήσουμε κάποιες ε, ιδέες σχετικά με το μέλλον του Urban. Πέρα δηλαδή από την πολιτική για τη συνοχή. Λοιπόν, γιατί ενδιαφέρομαστε για τις πόλεις, γιατί μας απασχολούν οι πόλεις. Καταρχήν, τα τρία τέταρτα περίπου του ευρωπαϊκού πληθυσμού ζει σε αστικές περιοχές. Οι πόλεις αναγνωρίζονται ως ε, μοχλή ανάπτυξης και κέντρα καινοτομίας. Οι πόλεις όμως αντιμετωπίζουν και προβλήματα. Υπάρχουν διαφορές, αποκλήσεις, χάσματα, πολλώσεις, κοινωνικές πολλώσεις που αποδυναμώνουν την οικονομική θέση των πόλεων. Πολλές φορές οι πόλεις δεν συνδέονται επίσης με το περιφερειακό επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να κάνουμε κάτι για τη δημογραφική πρόκληση, για το κλίμα, για τις εφοδιαστικές αλυσίδες, για την μετανάστευση και ούτω καθεξής. Η τρέχουσα οικονομική κρίση επιδεινώνει την θέση πολλών πόλεων, πολλών δήμων συγκεκριμένα. Αν δούμε την αστική διάσταση της τρέχουσας προγραμματικής περίοδου παρατηρούμε ότι καταρχήν διακόπηκε η λεγόμενη Community Initiative του Urban το άρθρο 8 του κανονισμού την αρίστοιχη μεθοδολογία την εφαρμόζουμε τώρα πλέον σε όλες τις πόλεις και όλες τις περιφέρειες. Θεωρητικά λοιπόν όλες οι πόλεις είναι επιλέξιμες για την χορήγηση ενίσχυσης για τους σκοπούς της συνοχής. Δεν χρησιμοποίησαν ε, το άρθρο αυτό όλες οι πόλεις βεβαίω. Βλέπουμε και αυτό είναι το θετικό της ενσωμάτωσης των μέρους μεθόδων σε μία είναι ότι το Urban ενσωματώνεται στα επιχειρησιακά προγράμματα με τρόπο αποδοτικό. Έχουμε περισσότερους πόρους στη διάθεσή μα, 10 δισεκατομμύρια. Και έχουμε επίσης και ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο, το Jessica, το οποίο ξεκίνησε με αργούς ρυθμούς, αλλά τώρα η λειτουργία του έχει επιταχυνθεί. Οι αδυναμίες μας παρατηρήσαμε ότι σε πολλά επιχειρησιακά προγράμματα η προσέγγιση ήταν τομεακή, στενά τομεακή. Δεν ήταν ενοποιημένη αν θέλετε. Οι πόλη σε τοπικό επίπεδο σε μικρό βαθμό και μόνο ανεπλάκησαν και δυστυχώς δεν αξιοποιήθηκε η πείρα που ανέφερε ο συνάδελφος προηγουμένως από την Community Initiative του Urban. Αν δούμε τώρα πώς εμπλέκονται οι τοπικοί πρωταγωνιστές, οι πόλεις αν θέλετε στο πρόγραμμα, στα διάφορα κρατημέλη, παρατηρούμε ότι εν γέννη η συμμετοχή είναι ανεπαρκής στον σχεδιασμό και στην ταύτιση στη συμμετοχή με τις δράσεις. σε πολλές περιπτώσεις η συμμετοχή περιορίστηκε στα τυπικά στην τυπική συμμετοχή κατά τη διάρκεια του αρχικού προγραμματισμού και όχι κατά τη διάρκεια της υλοποίησης. Οπότε οι περισσότερες πόλεις λοιπόν δεν συμμετείχαν καθόλου καν στη σχέση, στην φάση του προγραμματισμού. Τα προγράμματα όμως αυτά για να πετύχουν χρειάζονται, χρειάζεται να τα αγκαλιάσουν οι πόλεις αυτή είναι ακριβώς την αίσθηση της, της ταύτισης ε, με το έργο, πρέπει να την ενισχύσουμε. Το πρόγραμμα είναι φιλόδοξο, αναγνωρίζει τον ρόλο των πόλεων, στην επίτευξη των στόχων του 2020 όχι μόνο για την ε, εφορική ανάπτυξη αλλά για την ευφυή ανάπτυξη συνεπώς υπογραμμίζουμε σε κάθε περίπτωση ότι οι πόλεις πρέπει να συμμετάσχουν μετά στην έκθεση για τη συνοχή υπογραμμίζουμε ότι χρειάζεται οι πόλεις να συμμετέχουν περισσότερο στην υλοποίηση ε, να συμμετέχουν περισσότερο στις επιτροπές παρακολούθησης. Και η έκθεση για τη συνοχή καλεί επίσης τους εμπλεκόμενους να εθωρήσουν μια πιο ευέλικτη προσέγγιση στις περιοχές λαμβάνοντας υπόψη την γεωγραφική συνοχή. Είτε πρόκειται λοιπόν για μια γειτονιά, μια περιφέρει τη μια λεκάνη ποταμού. Αυτό χρειαζόμαστε. Η πρότασή μας επίσης λέει ότι πρέπει οι δράση να είναι σαφώς στοχευμένες υπέρ των περιοχών και των τομέων που βρίσκονται σε πλέον δινή θέση. Εκεί πρέπει να επικεντρώσουμε όλα τα θετικά στοιχεία της πρωτοβουλία. εκεί δηλαδή τα μέτρα να ενταθούν με τρόπο ενοποιημένο και με τρόπο που να εμπλέκει περισσότερο τους τοπικούς παράγοντες. Από τη φάση προς τα πάνω δηλαδή ε, χρειάζεται περισσότερη διαδικτύωση, περισσότερη δικτύωση μάλλον, αξιοποίηση του Urbact και βεβαίως να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τα χρηματοδοτικά μέσα για την αναγέννηση των πόλεων χάρη και στην εμπειρία από τον Τζέσικα. Ο Επίτροπος ενδιαφέρεται πολύ επίσης για μια ευρύτερη περιφερειακή ατζέντα, όχι μόνο για τη συνοχή, πέρα από τη συνοχή. Προσπαθεί να προωθήσει μια γενικότερη ανοιχτή συζήτηση, έναν διάλογο, ο οποίος θα μας επιτρέψει να κατανοήσουμε καλύτερα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι πόλεις. Ε, να δούμε αν υπάρχουν καλά παραδείγματα, καλές πρακτικές, πώς και τι πέτυχαν κάποιες πόλεις και πώς θα μπορούσε η πολιτική συνοχή να συμβάλλει στην ανηγέννη προσπάθεια. Η Γενική Διεύθυνση Ρέτζιο αυτή τη στιγμή τρέχει το πρόγραμμα Πόλης του Αύριο, Cities of Tomorrow. Στο πλαίσιο αυτό Οργανώσαμε ήδη δύο εργαστήρια. Ετοιμάζουμε και ένα τρίτο. Θα δημοσιεύσουμε φυσικά τα αποτελέσματα όλων αυτών των εργαστηρίων στο διαδίκτυο για να τα διαβάσετε. Η έκθεση πάνω στα είναι έτοιμη του χρόνου τον Μάρτιο και με πολύ χαρά θα συζητήσουμε και με την Επιτροπή σας τα αποτελέσματα του προγράμματος. Ο Επίτροπος επίσης υποστηρίζει την ε, εμπλοκή των ε, κρατών μελών και διαφορών ενώσεων το δίκτυο των αεφορικών πόλεων για παράδειγμα πρόκειται για ένα πρακτικό εργαλείο που θα βοηθήσει τις πόλεις να υλοποιήσουν τις αρχές του χάρτη της λειψίας για την εφορία. Η Γαλλία, το CMR και η Βελική Προεδρία και φυσικά η γενική μας διεύθυνση παρέχουν τεχνική υποστήριξη. Αυτή τη στιγμή ξεκινούμε την δοκιμαστική φάση σε 60 επιλεγμένες ευρωπαϊκές πόλεις η οποία θα κρατήσει ένα χρόνο. Ελπίζουμε μάλιστα ότι θα έχουμε θετικά αποτελέσματα τα οποία εννοείται θα είναι στη διάθεση όλων των ευρωπαϊκών πόλεων που επιθυμούν να τα χρησιμοποιήσουν, να τα αξιοποιήσουν. Αυτή είναι η τελευταία μου διαφάνεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον επόμενο μιλητή, τον κύριο Πολμπεβάν, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας του Eurocities. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε τρία σημεία στα πλαίσια του χρόνου που έχω στη διάθεσή την αρχή τη ολοκληρωμένη προσέγγιση. τη φιλόδοξη ε, αστική, στρατηγική ατζέντα που αναφέρθηκε και το θέμα της μεταβλητής γεωγραφίας. Νομίζω ότι οι αποδείξεις που είχαμε από το Ερμπάν ε, και τα δικά μας αποδικά στοιχεία μας οδηγούν στο να αναγνωρίσουμε ότι η πολιτική συνοχή έχει μεγαλύτερο και μακρύτερο αντίκτυπο ε, όταν ε, συνδυάζουμε περιβαλλοντικά και κοινωνικά μέτρα και υπάρχουν περιπτώσεις ε, όπου αυτή η ολοκληρωμένη προσέγγιση διεξάγεται καλύτερα, υλοποιείται καλύτερα σε τοπικό επίπεδο στις πόλεις. Το τοπικό επίπεδο είναι το επίπεδο που είναι πιο κοντά ε, στις συγκεκριμένες τοποθεσίες και οι πόλεις είναι αυτές που μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα τις πολιτικές αυτές και οι, οι πόλεις, το επίπεδο των πόλεων είναι το καλύτερο επίπεδο διακυβέρνησης και διαχείρισης. Έτσι λοιπόν, εκεί λειτουργούν καλύτερα τα πράγματα. Ξέρουμε ότι έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και ε, έχουμε καλύτερη αξία για τα χρήματα μας από μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Μόλις ακούσαμε ότι η ολοκληρωμένη προσέγγιση δεν έχει εφαρμοστεί ευρέως ε, στις ε, σημερινές στα πλαίσια των σημερινών δημοσιονομικών προοπτικών στο μέλλον πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο συντονισμό των προγραμμάτων ε, ε, μας ε, επιτρέπει να υλοποιήσουμε τα προγράμματα αυτά και φέτος το έτος για την καταπολέμηση της στόχιας μας δείχνει την ισχύ αυτής της ολοκληρωμένης προσέγγισης. Πρέπει να δούμε πώς διασυνδέεται η κοινωνική έντοξη με το ψηφιακό θεματολόγιο, με την κατάρτιση, την απασχόληση, καθώς ε, και την παροχή ποιοτικών κοινωνικών υπηρεσιών. Οι πόλει, άλλωστε, είναι συστήματα κοινωνική κινητικότητας. Ε, παρέχουν τις ευκαιρίες για την αύξηση των δεξιοτήτων, την αύξηση της ποιότητας ζωής, την αύξηση εργασίας, ε, συνεχώς ε, ανανεώνεται ο πληθυσμός της πόλης και αυτή η αστικοποίηση τελικά είναι τεράστια μηχανή παγκοσμίω. Και δεν πρέπει να ξεχνούμε το ρόλο των πόλεων ως ατμομηχανές της οικονομίας και της ανάπτυξης. Ε, το ευρωπαϊκό αστικό μοντέλο είναι ξεχωριστό. Έχουμε την ε, δυνατότητα ε, να έχουμε φόρους πόλεις που προσφέρουν καλή ποιότητα ζωής, καλές αστικές υπηρεσίες ξεχωριστές στην Ευρώπη, γιατί ε, ο τρόπος που γίνεται η αστικοποίηση στην Ευρώπη μας ε, θέτει σε θέση πρωτοπορίας εναντί ε, στον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό είναι κάτι που το υποστηρίζουμε. Αυτό το ευρωπαϊκό αστικό μοντέλο είναι κάτι που το υποστηρίζουμε και το προστατεύουμε μέσω των πολιτικών συνοχής. Είμαστε λοιπόν ικανοποιημένοι που βλέπουμε τη φιλοδοξία ατζέντα του Urban να ε, περιγράφεται στην πέμπτη έκθεση συνοχή, γιατί πιστεύουμε ότι η πολιτική συνοχή έχει να κάνει με το να ξεδιπλώνει την ε, ε, δυναμική, την εδαφική. Έτσι εμείς κατανοούμε την εδαφική συνοχή. Στα... Περάσαμε πάρα πολύ καιρό ε, στο πλαίσιο της χάραξης της πολιτικής συνοχής μιλώντας ε, για τη μείωση των ε, εδαφικών ενισοτήτων. Όμως εδώ πρέπει να ενισχύσουμε τη δυναμική και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι δεν έχουν όλες οι περιφέρειες την ίδια δυναμική και τις ίδιες λειτουργίες. Δεν αναμένουμε οι παραμεθόρες περιοχές ή τα νησιά πρέπει τόσο χάρη να έχουν το ίδιο ΑΕΠ να κατακεφαλήν όσο οι μεγάλες πόλεις στην Ευρώπη. Ποτέ δεν θα μπορέσουμε να μειώσουμε τις αποκλήσεις ε, κατά να ΕΠ με τον τρόπο που προτείνεται ορισμένες φορές. Πρέπει να αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν διαφορές και πρέπει να επικεντρωθούμε στα αποτελέσματα, ιδίως σε αυτό το κρίσιμο περιβάλλον καθώς βρισκόμαστε και σε μια ιδιαίτερη οικονομική συγκυρία. Πρέπει λοιπόν να ξεδιπλώσουμε την εδαφική δυναμική και όπου μπορεί να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο και εμεί θεωρούμε ότι αυτό πρέπει να γίνει στις αστικές περιοχές, το να ενδυναμώσουμε τα προγράμματα προκειμένου να τονίζονται τα αστικά ζητήματα με συγκεκριμένη κατανομή πόρων είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα μπρος και πιστεύουμε ότι πρέπει να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα και τα αποτελέσματα ε, επικεντρωνόμενοι εκεί όπου μπορεί να υπάρχει ο μεγαλύτερος αντίκτυπος, εκεί όπου ζει πλειονότητα των ατόμων, εκεί όπου οι επιχειρήσεις έχουν τη μεγαλύτερη εμπορική δυναμική, που έχουν αγορές και υπάρχουν δυνατότητες έρευνες και κοινοτομίας. Οι πόλεις πρέπει να είναι επικεφαλής της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας επίσης. Ε, ξέρουμε ότι και στις πόλεις παράγεται το 80% των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο των θερμοκηπίων στις ε, πόλεις. Ε, ο κοινωνικός αποκλεισμός και η φτώχεια είναι τα πιο μεγάλα προβλήματα. Αυτός είναι ένα μεγάλο στόχος ε, για την στρατηγική της Ευρώπης του 2020 η πρόταση της έκθεσης συνοχής ότι θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερο ρόλο στις αστικές αρχές κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή των αστικών στρατηγικών είναι ζωτική σημασία. Ακούσαμε από την Κομισιόν την αξιολόγηση Τη σημερινή κατάσταση. Ε, οι σημερινέ προοπτικέ είναι ότι οι αστικέ αρχές δεν εμπλέκονται. Συχνά υπάρχουν ε, συγκρούσει μεταξύ εντολών και εφαρμογή πολιτικών σε αστικό επίπεδο. Πρέπει λοιπόν να καταστήσουμε επιχειρησιακή αυτή τη φιλόδοξη αστική ατζέντα και στρατηγική. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι δεν ε, θα παραβλέπουμε περαιτέρω την αστική πτυχή. Ένα τμήμα, πρέπει να δίνουμε τμήμα των κονδυλίων ε, για την αστική ανάπτυξη, για την εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Θα πρέπει να έχουμε ένα σαφή σαφή κατάλογο ε, πόλεων ε, που θα ε, έχει καθοριστεί για κάθε κράτος μέλος σε συμφωνία με την Κομισιόν. Και τώρα έρχομαι στη μεταβλητή γεωγραφία. Ε, πέρα από αυτή την ε, διατομική προσέγγιση, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη έχει να κάνει και με την εδαφική ολοκλήρωση και υποστηρίζουμε να επιτρέψουμε μεγαλύτερη ευελιξία στην οργάνωση των επιχειρησιακών προγραμμάτων έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν καλύτερα την πραγματική γεωγραφία των ε, αναπτυξιακών διαδικασιών. Εμείς ε, θέλουμε να υποστηρίξουμε τη μεταβλητική γεωγραφία και ε, να δούμε πώς οι πόλεις στο επίκεντρο διάφορων περιοχών θα αποτελέσουν ε, ατμομηχανές της ανάπτυξης γιατί πρέπει οι πόλεις ε, να αναλάβουν ένα ρόλο και σε εδαφικό επίπεδο αλλά και σε διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος που προτείνουμε ναι, να αντιμετωπίσουμε τις σχέσεις μεταξύ αστικών κέντρων και υπαίθρου, δηλαδή να μην ε, προσπαθήσουμε να έχουμε ξεχωριστά προγράμματα ε, για την υπαίθρο και ξεχωριστά προγράμματα για τις πόλεις, αλλά κοινά προγράμματα. Θεωρώ ότι ε, αυτή τη στιγμή υπάρχει επίγουσα ανάγκη η Ευρώπη να έλθει σε πιο στενή σχέση με τους πολίτες τη και να επικεντρώσει τους πόρους και τις προσπαθήσεις της εκεί όπου ζει η πλειονότητα των πολιτών. Και αυτό και το επίπεδο διακυβέρνησης των πόλεων ε, είναι το καλύτερο. Είναι πολύ καλή ευκαιρία για μας για το μέλλον. Ε, ευφυής αηφόρος και συμμετοχική ανάπτυξη θα πετύχει στην Ευρώπη μόνο αν έχουμε ευφυείς αηφόρους και ε, συμπεριληπτικές πόλεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ενδιαφέρουσα σχόλιά σας κύριε Πολυμπεβάν και τώρα θέλω να δώσω το λόγο στον καθηγητή Λούντεξ Σίγκορα από το Πανεπιστήμιο Τσάρλς της Πράγας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Για να συζητήσουμε το, η θέση των Ευρωπαϊκών Πόλεων και Αστικών Κέντρων στην, στην Ευρωπαϊκή Πολιτική, θέτω τρία ε, ερωτήματα. Ποιος είναι ο ρόλος ε, στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, Κοινωνία. Ε, Ποιε είναι οι συνθήκες που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις οι πόλεις και ποιο είναι ο ρόλο τη πολιτική συνοχή στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων στην Ευρώπη. Θα μιλήσω για τις, μικρές και με, τις μεγάλες και τις μεσαίες πόλεις και θα σας δώσω την εμπειρία της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης ε, και των ε, νέων ε, κρατών μελών. Νομίζω ότι οι κοινωνίες του ΕΡΠΑ, οι αστικές κοινωνίες μάλλον, έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα εκ μέρους όλης της κοινωνίας. Είναι μεγάλες οι προκλήσεις και βασικές οι αντιδράσεις που χρειάζονται Πολύ συχνά ξεχνάμε τις ειδικότερε ε, αστικές ιδιότητες και συνθήκες που μπορεί να ισχύουν. Πάντοτε μιλάμε για το αν είναι διαθέσιμα τα κονδύλια. Από την άλλη πρέπει να ξέρουμε ότι για τις δράσεις χρειαζόμαστε εξωτερική χρηματοδότηση η οποία θα επιτευχθεί καλύτερα με την καλύτερη ενδογενή οργάνωση των πόρων. Έτσι λοιπόν ε, είναι πολύ μεγάλη ανάγκη ε, βιώσιμης ε, ανάπτυξης μιας κοινωνίας με οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική δυνατότητα επιλογών. Θα σας δείξω ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις και οι απαντήσεις που δίνονται σε αυτές στις πόλεις μας. Μία από τις βασικές προκλήσεις είναι η θέση των ευρωπαϊκών πόλεων στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα ε, σε σχέση πάντοτε και με τη γύρανση του πληθυσμού, το δημογραφικό πρόβλημα. Η απάντηση είναι να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών πόλεων και την ενεργό γύρανση. Δηλαδή να εμπλέξουμε όχι μόνο τους νέους αλλά και τους γυρότερους στην οικονομία. Ε, θα ενισχύσουμε έτσι την, την θέση μας. Επίσης, οι πόλεις πρέπει να χτίζονται γύρω από τις υπηρεσίες, την έρευνα και την ανάπτυξη, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση, έτσι ώστε να έχουμε ευρωπαϊκές πόλεις ε, οι οποίοι ε, θα εκμεταλλεύονται αυτό το κεφάλαιο. Να τονίσω το ρόλο της εκπαίδευσης. Τώρα με την οικονομική κρίση αυτό που κάνουμε συνήθως είναι να κόβουμε χρήματα από την εκπαίδευση. Νομίζω όμως ότι το βασικό μας περιουσιακό στοιχείο είναι οι άνθρωποι. Ο μορφωμένος πληθυσμός, η μορφωμένη οικονομία έχει επιλογές. Έτσι λοιπόν ε, μπορεί, μπορεί η έρευνα, η ανάπτυξη και η εκπαίδευση να είναι στόχοι, αλλά από την άλλη υπάρχουν και κάποια άλλα στοιχεία όπως οι καλύτερες μεταφορές, ε, τεχνολογίες πληροφοριών, ένα καλό περιβάλλον εργασίας που παίζουν και αυτά ρόλο. Δεύτερο επίπεδο που διάλεξα είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και ε, πόλεις με ενεργειακή αποδοτικότητα. Υπάρχει όλο και, αυξημένο κόστος, όλο και πιο αυξημένο κόστος ενέργειας και υπάρχει και θέμα ε, αποδοτικότητας ενεργειακής. Ένα λοιπόν από τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε είναι να φτιάξουμε ένα δομημένο περιβάλλον που θα έχει αποδοτικότητα σε επίπεδο ενέργειας και να οργανώσουμε την αστική δομή με βιώσιμο τρόπο. Να επικεντρωθούμε σε ένα περιφερειακό ε, μεταβατικό σύστημα το οποίο θα βοηθήσει την αστική επέκταση γύρω από τις πόλεις στην πετέρει περιοχή. Το τρίτο παράδειγμα που επέλεξα είναι η ανάπτυξη με συμπερίληψη των ανθρώπων. Πρέπει να φτιάξουμε πόλεις με επιπλογές οι πόλεις έχουν μεγάλη πολιτιστική και κοινωνική διαφοροποίηση και πολλές φορές χρησιμοποιούνται όροι όπως ε, διακρίσεις. Βλέπουμε ότι μειώνεται ο ρόλος της μέσης τάξης, ότι είναι μικτές, ε, δεν είναι πια μικτές οι κοινωνίες, αλλά υπάρχουν γετοποιημένες περιοχές και εκεί κάνω την έρευνά μου. Έτσι η κοινωνική ενσωμάτωση, η πολιτιστική ενίσχυση είναι πράγματα που ενισχύουν τη συνοχή με βάση την εκπαίδευση ε, και δεν, μιλάμε, δεν έχουμε μιλήσει πολύ για τους μικρο, με, μεσαίους. Αυτοί είναι που ουσιαστικά ε, οθούν την οικονομία και αυτοί είναι που θα πρέπει να συμμετάσχουν στην ολοκλήρωση. Πολλές φορές στις πόλεις μας οι πολιτικές ενσωμάτωσης και ολοκλήρωσης ε, δεν έχουν να κάνουν με κανονική ενσωμάτωση, αλλά με αφομοίωση. Έτσι λοιπόν, όταν μιλάμε για ενσωμάτωση, μιλάμε για μία ολοκλήρωση των ε, αστικών και μοιαστικών περιοχών, ενσωμάτωση κοινωνιών ε, διευρωπαϊκών. Χρειαζόμαστε καλύτερη λοιπόν υποδομές, ε, για μεταφορές, τεχνολογίες των πληροφοριών και καλύτερη προσβασιμότητα για να το πετύχουμε αυτό. Στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό των αστικών περιοχών έχουμε πετύχει πολλά στην αναδόμηση των ειστερημένων περιοχών, των ειστερημένων περιοχών. μιλάμε για μια ολοκληρωμένη και ισορροπημένη ανάπτυξη της πόλης στο σύνολό της, ενσωμάτωση των περιοχών, των προβληματικών περιοχών στην πόλη, Επίσης, ε, δικτύωση, ε, μιλάμε για την πολυκεντρική πόλη, πολυκεντρικά δίκτυα μέσα στις πόλεις, μεσαίου μεγέθους πόλεις, οι οποίες μπορούν να ε, μοιράζονται τις επιλογές και το δυναμικό της ευρύτερης αστικής περιοχής και μιλάμε και για τα διευρωπε... διεθνικά δίκτυα τα οποία ε, ε, έδειξαν ως τώρα από την εμπειρία μου τουλάχιστον ότι πιο πολύ κοιτάμε προς τις Βρυξές και το Λονδίνο παρά να ενισχύουμε τη συνεργασία μεταξύ των πόλεων. Άλλο θέμα είναι η συνέργεια, η σε επίπεδο οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών ε, στόχων. Η αρισιμότητα της ε, υποστήριξης είναι ένας από τους γενικότερους στόχους που έχουμε σε επίπεδο, για παράδειγμα, ενεργειακής αποδοτικότητας, η οποία πρέπει να είναι ένα δεδομένο, θα πρέπει να είναι δεδομένο στις ε, πολιτικές μας. Πρέπει να ενσωματώνουμε τους στόχους της έξυπνης, βιώσιμης ε, ανάπτυξης που σε περιλαμβάνει, που δεν ενισχύει τον κοινωνικό αποκλεισμό. Μιλήσαμε για πολυκεντρικές ε, περιοχές, ε, δίκτυο πόλεων, διεθνικές περιοχές. Νομίζω ότι πρέπει να εξετάσουμε την ευαίσθητη πλευρά της επικορικότητας και να δούμε πώς θα γίνεται η ίδια δράση συντονισμένα σε όλα τα επίπεδα ευρωπαϊκό, περιφερειακό και τοπικό. Τελική διαφάνεια παρακαλώ. Θα ήθελα οι πόλεις μας να είναι ανθεκτικές ή να είναι πόλεις οι οποίες μπορούν να αντιμετωπίσουν τις αβεβαιότητες που, ε, με τις οποίες ερχόμαστε αντιμέτωποι στο παρόν. Ε, πρέπει να υπάρχει ευελιξία στη διαχείριση, να συμφιλιώνονται οι ειδικοί στόχοι με τους γενικότερους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα με τις συνθήκες της συγκεκριμένης κάθε πόλης. Χρειάζεται λοιπόν μια προσέγγιση η οποία θα ενισχύσει την ενδογενή ανάπτυξη του περιβάλλοντος και έτσι θα έχουμε τη δυνατότητα πειραματισμού, ανατομίας ε, και δικτύωση μεταξύ των πόλων. Αυτό λοιπόν που προτείνω είναι καλύτερη, μεγαλύτερη διακριτικότητα σε τοπικό περιφερειακό επίπεδο ε, που θα αντικατοπτρίζει ε, τις αστικές και περιφερειακές συνθήκες μέσα στα πλαίσια της, αντι... της των ευρωπαϊκών στόχων. Ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά για την ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας. Ε, τώρα δίνω το λόγο στον επόμενο ομιλητή, Ευχαριστώ πολύ. Έχω εξεδησει κατά αρχή, ότι Ιβαν Τόσιξε του Μετροπολιτικού Ερευνητικού Ινστιτούτου της Βουδαπέστης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Έχω έξι δηλώσει καταρχήν ότι η στρατηγική για την, ε, το 2020 είναι ένα καλό σημείο αφετηρίας ε, για τη μελλοντική πολιτική συνοχής η περιβαλλοντική φορεία και το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο θα πρέπει να συνοδευτούν από τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη. Όμως δεν είναι εύκολο να επιδεχθούν οι στόχοι αυτοί για την αντιφατική μεταξύ τους ε, και κάθε πολιτική που θα επιδιώκει τον ένα στόχο θα δημιουργεί προβλήματα στου υπόλοιπου στόχου ή μονοπλευρή ε, έμφαση στην οικονομική αποδοτικότητα μπορεί να οδηγήσει σε απειλητικά ε, παραδείγματα πόλεων που θα μείνουν πίσω, που θα υστερούν. Είδαμε τέτοιες περιπτώσει στι Ηνωμένες Πολιτείες και στο οικονομικοί στόχοι για το 2020 θα μπορούσαν ε, να βελτιωθούν ε, αν ε, αυξήσουμε και το ρόλο των περιαστικών περιοχών. Ε, θα πρέπει να εξαρθούν οικονομικά μέσα για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συμπεριλήψη. Οι ε, νέε κατασκευέ ε, με μηδέν εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα είναι πολύ πιο ακριβέ από ότι η ανακαίνιση των υφιστάμενων κατοικιών και επίσης ε, η συγκέντρωση μπορεί να οδηγήσει τους πλουσίους να κατελείψουν τις πόλεις. Σας δώσω ένα παράδειγμα, εδώ βλέπετε ε, μία πόλη πολύ πυκνοκατοικημένη, αυξάνεται η πυκνότητα μέσα στην πόλη και αρχίζουν ε, να γκρεμίζουν κάποιες γειτονιές και φεύγουν οι φτωχοί για να γίνει ανάπλαση της πόλης, για να κατοικήσουν οι πλουσίοι. Έτσι λοιπόν κάτι τέτοιο μπορεί να είναι πολύ κακό για τους φτωχούς. Εδώ βλέπετε ένα άλλο παράδειγμα σε ένα από τα νέα ε, οι αποκλεισμένοι Ρωμά έχουν πολύ καλύτερε συνδικέ εργασίας, αλλά 20 ε, χιλιόμετρα ε, μακριά από την πόλη, η επένδυση αυτή οδηγήθησε στο να αποκλειστούν εντελώ από την κοινωνία. Η πολιτική συνοχή είναι μεγάλη πολιτική αναπτυξιακή και ε, πρέπει να οδηγήσει σε ε, καλές επιδόσεις, γιατί οι μεγάλες περιοχές μπορούν να συνεισφέρουν στην Ευρώπη και επίση είναι πολύ σημαντικό ε, να πληρωθούν οι στόχοι του 2020 με έναν ολιστικό τρόπο. Ε, ο προπολογισμό για την πολιτική συνοχή θα πρέπει να διατηρηθεί τουλάχιστον στο σημερινό επίπεδο και μια ισχυρή πανευρωπαϊκή πολιτική συνοχής ε, χρειάζεται με ιδιαίτερη έμφαση στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη για να ε, καταπολεμηθούν εξωτερικοί παράγοντες. Εδώ βλέπετε πως το 1936 είχαν χαραχθεί οι αυτοκινητρόδρομοι στην Ευρώπη. Τότε δεν υπήρχε ακόμη ε, το ε, σιδηρούν παραπέτασμα. Το 1945 δημιουργήθηκε και τι έγινε μέχρι το 1996. Τίποτα δεν έχει γίνει στα νέα κρατημέλη, ενώ πολύ περισσότεροι αυτοκινητοδρόμοι έχουν κατασκευαστεί στην Δυτική Ευρώπη. Έτσι λοιπόν σημαίνει ότι πρέπει να ε, διοχετεύσουμε πόρους και στα νέα κράτη-μέλη. Τώρα, πώς ε, ε, λειτουργεί με ένα ολοκληρωμένο τρόπο η πολιτική συνοχή. Ε, μπορούμε να διασφαλίσουμε τους στόχους του 2020 στην εφαρμογή στις πόλεις, στις περιφέρειες, σε τοπικό επίπεδο. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε ταυτόχρονα τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές πολιτικές. Πρέπει να πολεμήσουμε τον αποκλεισμό των μεταναστών ε, και των ε, μειονοτικών πληθυσμών. Ε, όμως δυστυχώς σε ό,τι αφορά τη διοικητική σκοπιά είναι αδύναμες οι πόλεις. Μπορούμε να πούμε ότι η Ευρώπη έχει εδαφικά συστήματα του 19ου αιώνα. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει, θα πρέπει να δοθούν κίνητρα προκειμένου να έχουμε καινοτόμε εξελίξεις. Εδώ βλέπετε ένα παράδειγμα στη Βουδαπέστη όπου η η πόλη είναι το κίτρινο κομμάτι, θα πρέπει να συνεργαστεί με τις ε, γειτονικές πόλεις, αλλά αυτή στη στιγμή είναι πολύ αδύναμη συνεργασία. Ποια πρέπει να είναι τώρα η αστική διάσταση της πολιτικής συνοχής. Νομίζω ότι το πνεύμα του Urban πρέπει να επανέλθει, αλλά ε, όχι με τη μορφή του Urban 3, γιατί το Urban είχε πάρα πολλές αδυναμίες. Ε, ε, ουσιαστικά δεν έδωσε τίποτα στις όμορες περιφέρειες και δεν ασχολήθηκε με τις κύριες αιτίε για την καταπολέμηση της στόχιας. Πολλοί είπαν ότι οι παρεμβάσεις σε μικρές περιφέρειες απλώς είχαν ε, να κάνουν ε, με ε, κάποιες παρεμβάσεις παραδείγματος χάρη όπως ε, να φτιάχνουν τις καρέκλες όταν ο Τιτανικός βυθίζεται. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει ολοκληρωμένη προσέγγιση σε ευρύτερες αστικές περιοχές για να αποφευχθεί προσπαθούν οι πρόσθετες μελλοντικέ τομεικέ πολιτικές και πρέπει φυσικά να έχουμε το κατά νου και την απασχόληση. Εδώ βλέπετε ένα παράδειγμα μιας μη ολοκληρωμένη ε, προσέγγισης, 20 ε, χιλιόμετρα από ε, το κέντρο της πόλης, η Ευρώπη πρέπει να παίξει ισχυρό ρόλο για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό, γιατί οι αποφάσεις σε εθνικό επίπεδο δεν είναι πάντα προς αυτή την κατεύθυνση. Φυσικά δεν υπάρχει μία λύση που να ταιριάζει σε όλους, διαφορετικές πολιτικές έχουν ε, διαφορετικό εδαφικό πεδίο. Όμως πρέπει να υπάρχει επαρκή ευελιξία, να περιγραφούν οι ελάχιστες προϋποθέσεις για την ε, ολοκληρωσή και να πετύχουμε τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει και επαρκή συμμετοχή των ενδιαφερομένων. Θα έλεγα λοιπόν ε, ότι ε, το ουγγρικό αναπτυξιακό σχέδιο αποτελεί πραγματική επιτυχία ολοκληρωμένου σχεδιασμού ως ερεσιμότητα για ως όρο για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, πρέπει, στην περίπτωση, για να λάβουμε τα χρήματα πρέπει να έχει υπογραφεί και από εθνικούς εμπειρογνώμονες ε, το σχέδιο. Ε, θα ε, πρέπει επίσης να ακολουθήσουμε έναν τρόπο, έναν, μια μέθοδο από τη βάση, από κάτω προς τα πάνω. Οι στρατηγικές ανάπτυξης θα πρέπει να επικεντρώνουν όλους τους ευρωπαϊκούς πόρους και από το Κοινωνικό Ταμείο και από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ε, κανένα project δεν πρέπει να λαμβάνει κοινωτική χρηματοδότηση αν δεν έχει εγκριθεί στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης εδαφικής αναπτυξιακής στρατηγικής της ε, και, ε, και αν δεν συνδέεται με την επίτευξη των στόχων του 2020 και όλες οι συναλλακτικές ιδέες όπως ε, ε, τα αστικά αναπτυξιακά ταμεία θα πρέπει να υπόκειται στα ολοκληρωμένα αναπτυξιακά εργαλεία. Εδώ βλέπετε πέντε επιλογές. Οι πρώτες δύο είναι ισχυρέ επιλογές. Αν μπορούσαμε να έχουμε μία οδηγία για την οδηγία πλαίσιο για την και ανάπτυξη που θα έμοιαζε με την οδηγία που έχουμε για το ΙΔΟΡ. Ε, η δεύτερη επιλογή θα είναι να έχουμε ε, μία ερεσιμότητα ε, που είναι η ουγγρική προσέγγιση. Οι άλλε τρει είναι πιο αδύναμε επιλογέ, δεν θα τι πρότεινα. Η ανοιχτή μέθοδο είναι πάρα πολύ αδύναμη και η μέθοδο αναφορά επίση συμπεράσματα εδώ. Έχουμε τις έξι δηλώσεις, καλή φετηρία η στρατηγική το 2020, η πολιτική συνοχή πρέπει να έχει δει το στόχο και είναι σημαντική και η ολοκλήρωση, καθώς η πολιτική συνοχή πρέπει να επικεντρωθεί σε αστικές περιοχές και στη λειτουργία των αστικών περιοχών. Το πνεύμα του Urban θα πρέπει να επανέλθει, όχι το Urban 3 ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δυναματίσει ισχυρό ρόλο ε, για ε, την υλοποίηση ολοκληρωμένου σχεδιασμού, διαφορετικά δεν θα γίνει. Και τέλο, υπάρχουν τρόποι να δημιουργήσετε μια πολιτική συνοχή μετά το 2013 που να βασίζεται σε στρατηγικέ ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη και οι παρεμβάσει τη πόλη ε, δεν πρέπει να στοχεύουν στο να ομορφαίνουμε το δημόσιο χώρο, αλλά να βελτιώνουν και τη ζωή των πολιτών που χρησιμοποιούν το χώρο αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας. Ε, τώρα θα ήθελα να ζητήσω να ανάψουν τα φώτα για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Να δώσω στον Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να βγάλω τρία συμπεράσματα από όσα άκουσα. Το πρώτο είναι και χαίρομαι για το είπε ο καθηγητής ε, Τρόσκι ε, να δίνουμε ευρωπαϊκά κανδύλια μόνο όταν εμπλέκεται και η τοπική κοινωνία. Είναι ε, απαραίτητο να υπάρχει ε, στα διαχειριστικά προγράμματα ε, μια συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών. Αυτό είναι ανεπαρκές προς το παρόν και γι' αυτό είναι και ο λόγος που πολλά προγράμματα δεν ανταποκρίνονται στα, στις απαιτήσει. Ένα δεύτερο σημείο που θέλω να θέξω έδειξε και ο καθηγητής Ικόρης, είναι η, ενεργητική, η απόδοση της ενέργειας. Είναι φιλόδοξοι οι στόχοι που θέθηκαν στην Κοπενχάγη, όμως όταν μιλάμε για την πολιτική συνοχή θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες αστικές περιοχές όπου υπάρχουν κτίρια τα οποία χρειάζονται ανακαίνιση και ε, θα έχουν ε, τη δυνατότητα να κάνουν αυτή την ανακαίνιση μόνο αν δώσουν πολλά χρήματα παρόλο που δεν έχουν τόσα χρήματα οι φτωχές αυτές τις περιοχές. Αυτό είναι ένα στοιχείο, ε, η δυνατότητα των εφιστάμενων διαρθρωτικών ταμείων να δώσουν χρηματοδότηση για την εξυγίανση των ε, περιοχών, των γειτονιών που έχουν ανάγκη για ανακαίνιση των κτηρίων τους ε, και στις νέες χώρες αλλά σε όλα τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις όπου δεν θα υπάρχουν, για παράδειγμα, σκηνές ε, στη Γερμανία. Τέλος, καθηγητής Χειροσικόρα μίλησε για την μετανάστευση. Στη δική μου χώρα έχουμε σε όλες τις μεγάλες πόλεις το 50% των νέων κάτω των 18 ετών έχουν υπόβαθρο μεταναστευτικό και υπάρχει και μεγάλο ποσοστό του συνολικού πληθυσμού στην ε, περιοχή μου που έχει τέτοιο υπόβαθρο. Θεωρώ λοιπόν ότι τα διαρθρωτικά ταμεία όταν σκεφτόμαστε το 2020 και τη στρατηγική της Λιζαφώνα πρέπει τα ταμεία ε, να φτιάχνουν υποδομές και για την ενίσχυση αυτών των νεαρών ομάδων γιατί ε, αν σκεφτούμε ότι αυτός είναι ένας οικονομικός παράγοντας ο οποίος ε, ε, παραμένει αχρησιμοποιητός, οι άνθρωποι αυτοί δεν χρησιμοποιούνται, ε, όταν μιλάμε για προβλήματα δημογραφικής αλλαγής και τα λοιπά, θα μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Με οικονομική ενίσχυση λοιπόν, αν είμαστε πιο δραστήριοι μέσα σε αυτή την περίοδο. Ευχαριστούμε πολύ, Πίτερ. Επειδή έχουμε μισή ώρα, να ζητήσω από τους ε, πυρογνώμονες ε, να απαντήσουν σύντομα και μετά να δώσω στον ε, συνάδελφο Όλμπριχτ το λόγο. Ποιος θέλει να μιλήσει. I can give Μια σύντομη απάντηση για ένα σημείο. Το συμπέρασμά σας για την εξελόγηση το Urban 2, ναι, με βρίσκει σύμφωνο. Πρέπει να συμμετάσχει στην αξιολόγηση και η τοπική κοινότητα. Κάτι άλλο, σχόλιο. Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ. Συμφωνία. Κύριε Σόλμπριχτ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Στο πλαίσιο της συνοχής ε, η αστική διάσταση γίνεται όλο και πιο ενδιαφέρουσα. Αλλά θέλω να ρωτήσω τους ειδικού για κάποιες ειδικέ πτυχές. Μετά από την πέμπτη έκθεση έχω την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει χάσει τον ενθουσιασμό της για την εδαφική συνοχή. Και το είδα και το άκουσα στην ομιλία του κ. Τεγκράν. Δεν νομίζω ότι έχει περάσει η εποχή τη εδαφική συνοχή. Η ερώτησή μου λοιπόν προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πιστεύουμε ακόμη ότι η εδαφική συνοχή είναι πολύ σημαντική, παραμένει πολύ σημαντική. Το λέει φυσικά η συνθήκη, αλλά ε, πέραν αυτού. Το δεύτερο στοιχείο είναι γιατί γιατί η ένταξη της αστικής διάστασης στην πολιτική συνοχή απέτυχε. Γιατί απέτυχε. είναι εξαιρετική ιδέα. Γιατί δεν αποδίδει στην πράξη όμως η κίνηση αυτή. Είναι λόγω έλλειψης πολιτικής βούλησης, λόγω έλλειψης μηχανισμών, μέσων, μεθόδων. υποχρεώσεις για τα κράτη-μέλη ενδεχομένως όσον αφορά τις διαχειριστικές αρχές. Εγώ θα λέω ότι μάλλον αυτό συμβαίνει. Οπότε προς τον κύριο Τενέλη μου και η ερώτησή μου είναι ποια ήταν η οικονομική, η χρηματοδοτική συλλογιστική του προγράμματος. Δεν φταίει μόνο η πολιτική βούληση. Υπάρχουν τώρα εξαιρέσεις στο Περιφερειακό Ταμείο που δεν ίσχυαν για την λεγόμενη δισταυρούμενη χρηματοδότηση. Κάτι το οποίο έκανε πολύ δύσκολη την κατάσταση. Περιέπλεξε τα πράγματα ω προ το Urban. Εξηγήστε μου τι ακριβώ συνέβη. Γιατί στην αρχή αυτή τη σύσκεψη μιλάγαμε για συνέργειε. Πού πήγαν αυτέ οι συνέργειε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την πείρα που έχουμε από την συνδυασμένη χρηματοδότηση, δηλαδή μέσω των διαφορετικών ταμείων, για να πετύχουμε και εδώ. Γιατί οι διαχειριστικέ αρχέ, στο πλαίσιο κάθε ταμείου, έχουν την υποχρέωση να προβούν σε περικοπέ. Το ΕΠΕΝ όμως δεν δουλεύει με ένα μόνο ταμείο. Και πείτε μου λοιπόν. Και μετά από του δύο καθηγητές θέλω να πω το εξή. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά, αλλά υπάρχει στην ατζέντα του 2020 μια μη ρεαλιστική ιδέα ότι μπορούμε να πετύχουμε του στόχου. περί εφορία, ένταξη κλπ. ξεχωριστά. Το να αποκοπούν ο ένα από τον άλλον αυτοί οι στόχοι είναι μη ρεαλιστικό. Αποκλείται να πετύχουμε οτιδήποτε. οποίο το σχεδίασε νομίζω πρέπει να επανέλθει στην πραγματικότητα. Ευχαριστώ πολύ. Λέει πρόεδρος. Οι ειδικοί και πάλι έχουν να πούν κάτι. σχετικά με την εδαφική συνοχή. Πέρα τη συζήτηση για την πράσινη βίβλο, η κατάσταση έχει ως εξής. Τα κρατημέλη και οι άλλοι εμπλεκόμενοι είπαν ότι δεν έχουμε χρόνο να χάσουμε, πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα για την εδαφική συνοχή με βάση συγκεκριμένους στόχους, σε συγκεκριμένους τομείς ώστε η στρατηγική να αποκτήσει πιο συγκεκριμένη απτή διάσταση. Ένα, θα προσθέσουμε δηλαδή στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο και μια, ένα κεφάλαιο για την εδαφική συνοχή. Κατά δεύτερο λόγο, θα ζητήσουμε περισσότερη συνέπεια της πολιτικής συνοχής με την εδαφική διάσταση η Κομισιόν θα εντείνει τι προσπαθίε σε αυτόν τον τομέα και ξεκίνησαμε συναφώς διάλογο με τα κράτη-μέλη και τρίτον θα χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία που έχουμε αποκομίσει και πλέον θα λάβουμε υπόψη μας περισσότερο τις απαιτήσει ε, τις τοπικές των συγκεκριμένων πόλεων και προτείνουμε επίσης να υποστήριξουν περισσότερο την τοπική ανάπτυξη στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Αυτά είναι μερικά πρακτικά πράγματα από την πλευρά της Κομισιόν τα οποία λοιπόν χωρίς να περιμένουμε κάποιες άλλες μεγάλες ε, πρωτοβουλίες σε ανώτερο επίπεδο με ρώτησε κάποιο συγκεκριμένα για το πώ συνδυάζουμε τα ταμεία. Έχετε απολύτω δίκιο. Το Urban 2 ήταν 100% ευέλικτο. Μεταξύ, μπορούσε να διαλέξει δηλαδή μεταξύ μέτρων του Περιφερειακού και του Κοινωνικού Ταμείου. Αν και τα περισσότερα χρήματα ήρθαν από το Περιφερειακό, το πρόγραμμα είχε απόλυτη διακριτική ευχαίρεια για το πώ θα ξοδέψει τα χρήματα αυτά. Επρόκειτο περί μείγματο λοιπόν, όμω, ε, για παράδειγμα στο Μπόρι, στην ε, ε, Σουηδία τα χρήματα εξοδεύτηκαν σε προγράμματα κοινωνικά, εκπαίδευση. Ενώ το Μπραντεμπούργκ στην ε, Γερμανία ε, κινήθηκε με βάση μέτρα του Περιφερειακού τομείου Και φυσικά ισχύουν και όλε οι ενδιάμεσε λύσει. Άρα, αν δεν υπήρχε αυτή η ευελιξία, πραγματικά δεν βλέπω πώ θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει τόσο πολλά πράγματα. άλλο σχόλιο από του ειδικού, παρακαλώ. Γιατί ρώτησε κάποιο, δεν εντάσσει τη δευχή συνοχή και στη σημερινή προσέγγιση. Κοιτάξτε, υπάρχουν μερικέ εξαιρέσει. Δεν απέτυχε αυτή η υπόθεση και στι κατοχώρε έχουμε ένα παράδειγμα περιοχών και πόλεων που πέτυχαν. Μετά υπάρχει το Βερολίνο. Πάντως γενικά, όπως προείπα, εμείς που έχουμε δουλέψει σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο στα κράτη-μέλη, ξέρουμε ότι σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις. Ε, υπάρχουν προβλήματα, πολιτικοί ανταγωνισμοί, διαφορές και πολλές φορές στο περιφερειακό επίπεδο οι άνθρωποι ε, προσπαθούν να κάνουν τα πάντα με πεπερασμένους πόρους αποδυναμώντας τα μέτρα όμω σε τοπικό επίπεδο λόγω της περιορισμένης χρηματοδότησης και το ίδιο ισχύει και λόγω των αντικρουμένων ε, αναγκών και σε ένα ανώτερο επίπεδο. Τα κράτη-μέλη λοιπόν δεν έχουν αξιοποιήσει αυτή την εναρμόνιση του Urban. Ο στόχος πάντως είναι τα κονδύλια για το Urban να αξιοποιηθούν και ήταν καλή αυτή η εξέλιξη. Παρ' όλα αυτά κάποια περιφέρεια θα έχει πάντα τον πειρασμό να πει εγώ τις δράσεις του Έρμπαν θα τις ε, κατρίμω σε όλη μου την περιφέρεια ε, αντί να τα εστιάσω τα χρήματα αυτά εκεί που υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Γι' αυτό η Κομισιόν δεν έχει γράψει βεβαίως από αυτό, ε, το προτείνει ε, να υπάρχουν απευθείας διαπραγματεύσεις συγκεκριμένων πόλεων με τις κυβερνήσεις. Κυρία Δωσίκοφα. Δεν ε, ήθελα να δώσω τη λάθος εντύπωση μεταξύ της υφόρου βιώσιμης και συμμετοχικής ανάπτυξης. Εγώ ήθελα να πω ότι απλώς πρέπει όλα να εργάζονται ε, σε συνέργειες και όλα αυτά πρέπει να αποτελούν προϋπόθεση για την ε, υλοποίηση και την εφαρμογή αυτών των πολιτικών. Είχα τόσο λίγο, τόσο χρόνο που δεν μπορούσα να δώσω παραδείγματα αλλά θα αναφέρω ένα στε αυτές ε, τις πόλεις όπου μιλάμε για πολιτιστική και κοινωνική ένταξη. Η μεγαλύτερη ένταξη συμβαίνει στο χώρο εργασίας, αλλά και σε εκπαιδευτικά ιδρύματα όπου τα οποία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για αυτή την ένταξη και όταν μιλάμε για το ρόλο της εκπαίδευσης μπορούμε να μιλήσουμε για το ρόλο των πανεπιστημίων στις πόλεις έτσι ώστε να μιλάμε για σύνδεση της εφηούς ανάπτυξης με ε, την ανάπτυξη όπου μπορούν όλοι να συμμετέχουν και πρέπει να δούμε ότι τώρα χάνουμε αριθμό γιατί έχουμε ε, τώρα μικρότερε γενιέ ανθρώπων που έρχονται στο σχολείο και επίση ε, χάνουμε και ε, φοιτητέ γιατί φεύγουν στι ΗΠΑ ή φοιτητέ που από τις χώρες της Ανατολική Ευρώπης πηγαίνουν ε, στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Πρέπει να αποφύγουμε αυτή τη διαρροή. Πρέπει λοιπόν ε, να ε, έχουμε Κάποιε δυνατότητε ε, τέτοιε τη πόλη μα ώστε να αποφύγουμε αυτά τα αποτελέσματα. Και αυτό πρέπει να το συνδέουμε με του στόχου βιώσιμη ανάπτυξη, γιατί νομίζω ότι αν έχουμε καλά εκπαιδευμένο πληθυσμό, τότε έχουμε και καλύτερε ε, επιδόσεις και με καλύτερε δεξιότητε. και φυσικά έχουμε και ανθρώπου οι οποίοι θα συμπεριφερθούν και διαφορετικά και στον τρόπο τη ζωή του, θα δίνουν μεγαλύτερη προσοχή σε θέματα υφορία. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι ένα ολοκληρωμένο στόχο στόχους ανάπτυξης αυτών των τριών ε, στόχων. Ε, μιλάμε για μια ευφυή αηφόρο e ανάπτυξη με τη συμμετοχή όλων. Εγώ δεν έχω τόσο κακή άποψη για τη στρατηγική για το 2020 τουλάχιστον. Ε, σε αυτό το εγγραφό έχουν τεθεί πέντε συγκεκριμένοι στόχοι και ποτέ δεν έχω δει ε, σε άλλο έγγραφο στο παρελθόν ε, να τίθενται συγκεκριμένοι στόχοι σε κοινωνικό επίπεδο. Όμω θα πρέπει να τους συνδέσουμε αυτού του στόχου. και θα πρέπει να υπάρχει πραγματική συζήτηση στα πλαίσια των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων με τις πόλεις για να δούμε πώ μπορούν να υλοποιηθούν στόχοι αυτοί. Θα πρέπει και σε επίπεδο τοπικό ε, να γίνει προβληματισμός για το πώς ε, θα ε, δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, θα μειωθούν οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και πώς θα σκεφτούμε, το χάρη, να μην χτίσουμε νέα σπίτια για τους πλούσιους, αλλά να ανακαινήσουμε ε, τα υφιστάμενα κτίρια, γιατί κάτι τέτοιο θα βοηθήσει να μείνουν και επιτόπου οι άνθρωποι και να ξεπεράσουν τις οικονομικές δυσκολίες. Έτσι λοιπόν, ε, εγώ νομίζω ότι έτσι μπορούμε να υλοποιήσουμε αυτούς τους στόχους και να έχουμε και αυτούς τους ε, πέντε κύριους στόχους. Πριν δώσω το λόγο στην κυρία Ντελή, θα ήθελα να ρωτήσω αν θέλετε το λόγο για να απαντήσετε. Ναι, νομίζω ότι συνεννοούμαστε πολύ καλά μεταξύ μας, ε, κύριε Σίκορα. Ε, μου αποδείξατε με την παρέμβασή σας ότι υπάρχει ε, τάση και δεν πρέπει να το κρύβουμε ότι θα πρέπει να ε, έχουμε ε, τριμερείς ε, πολιτικές ευρωπαϊκές και δεν πρέπει ε, να κρύψουμε ότι η πολιτική συνοχής και η αστική διάσταση θα πρέπει να είναι κάτι που συμπεριλαμβάνει τους όλους. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να επικεντρωθούμε στους πέντε στόχους που εντάσσονται στη στρατηγική για το 2020 και να μην μιλάμε για κατακαιρματισμό γιατί μιλάμε για ολοκληρωμένη προσέγγιση και στην αναθεώρηση του προπολογισμού μία από τι δυνατότητε είναι να κατακαιρματίσουμε τον προπολογισμό σε διάφορα μέρη. Έτσι λοιπόν, ε, η αστική διάσταση μα δείχνει ότι δεν είναι ρεαλιστικό και είναι αδύνατο να γίνει κάτι τέτοιο. Και αυτό που είπε ε, ο καθηγητή ε, Μέρκετ, έχουμε πάρα πολύ σαφεί στόχου και πολύ ωραία συνθήματα. Και δεν θα πρέπει να κατακαιρματίσουμε τον προπολογισμό σύμφωνα με τα συνθήματα αυτά που έχουμε. Μάλιστα, σα ευχαριστώ πολύ. Κυρία Αντελή, ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να επανέλθω στην εξή διαπίστωση. Ότι τα κεκτημένα του Urban σήμερα έχουν ε, αποδυναμωθεί για να μην πούμε ότι έχουν χαθεί στο mainstreaming της ε, δραστικής πολιτική και τη πολιτική συνοχή, γιατί το Έρμπαν ε, είχε καταδείξει τρει ε, κύριε θετικέ πτυχέ. Ε, είχαμε την καλύτερη συνεργασία και το συνδυασμό μεταξύ των τομέων, ενίσχυση των πρωτοβουλειών με μια οριζόντια εταιρική σχέση σε τοπικό επίπεδο και συγκέντρωση των πόρων σε ε, συγκεκριμένες παρεμβάσεις που μας επέτρεψαν να έχουμε μια πραγματικά ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ανάπλαση των πόλεων, ενεργοποιώντας όλους τους πρωταγωνιστές και είχαμε παρέμβαση ε, όλων των τομέων. Έτσι λοιπόν, και είχαν καταστεί και υπεύθυνοι οι ε, τοπικοί παράγοντες. Έτσι λοιπόν μπορούσαμε να έχουμε εκεί με το Urban μια καινοτόμο προσέγγιση για την παρεμβάση Τη της και το urban δεν συνεχίστηκε στο mainstreaming ε, στη σημερινή προγραμματική περίοδο. Έτσι λοιπόν η δυνατότητα της ε, ε του πολλαπλησιασμού της συμμετοχής των πόλεων ε, δεν προωθείται, είναι ακόμη πάρα πολύ μακριά από τα επιχειρησιακά προγράμματα ε, γιατί ουσιαστικά αποτελούν ε, μόνο παραλήπτες των πολιτικών. Έτσι λοιπόν πρέπει να σκεφτούμε πώς στην επόμενη προγραμματική περίοδο θα επανεισαγάγουμε την ολοκληρωμένη προσέγγιση για την υλοποίηση ε, του Ερμπαν και πώς θα έχουμε έναν άξονα ε, πολιτικής συνοχής για την ανάπλαση των πόλεων έτσι ώστε στις πόλεις να ενεργοποιηθούν ε, οι αρμόδιοι φορείς για να παρέμβουν στις ε, συνοικίες ε, οι οποίες αντιμετωπίσουν δύσκολες συνθήκες. Μία ευρωπαϊκή χρηματοδότηση θα αποτελούσε ένα μοχλό για την ενεργοποίηση των επενδυτών με καινοτόμα χρηματοοικονομικά μέσα όπως είδαμε από το πρόγραμμα Jessica και αυτή είναι η πρώτη μου διαπίστωση. Ε, στη συνέχεια θέλω να αναφερθώ στις ε, κλιματικές προκλήσεις. Μπορώ να σας πω ότι είμαστε σε επιδακτική ε, κατάσταση. Η μάχη για το κλίμα και οι κλιματικές προκλήσεις ε, θα αντιμετωπιστούν στις πόλεις και σήμερα θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι πολιτικές διακυβέρνησης ε, στις πόλεις γιατί έχουμε ευθύνη. Δηλαδή πώς αύριο θα δημιουργήσουμε αϊφόρους πόλεις. Και όταν είναι αϊφόρες πόλεις, προσοχή. Δεν υπάρχει ένα προκαθορισμένο κουτί, ε, γιατί υπάρχουν διαφορές μεταξύ των ε, διάφορων επικρατιών. Ε, βρισκόμαστε εδώ σε μια στρατηγική για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και της μείωσης των εκπομπών, αλλά θα πρέπει όλα αυτά να τις σκεφτούμε εν ώψη της μελλοντικής αναγέννησης των πόλεων και σήμερα ε, οι κύριοι πρωταγωνιστές για τη μάχη αυτή είναι οι πόλεις. Το επαναλαμβάνω. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Ποιος εμπειρογνώμων θέλει να απαντήσει πρώτος. Ε, Συμφωνώ ότι το ε, πνεύμα της ενσωμάτωσης και ολοκλήρωση έχει χαθεί στο mainstreaming. Το θέμα είναι πώς θα το επαναφέρουμε. Είναι πάντοτε λάθος να επαναρχόμαστε στην ίδια διαδικασία, να βρίσκουμε 70 μέρη ε, στην ε, Ευρώπη που είναι σε παρακμή και εκεί πέρα να επικεντρώνουμε όλοι μας ε, τη δράση. Θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο ευρύς ε, στον τρόπο που σκεφτόμαστε. Η περιφέρεια, η πόλη, ευρύτερη να σκέφτεται ποια είναι τα σημεία που χρειάζεται καλύτερη παρέμβαση. Γιατί άλλες φορές είναι τα κτίρια, άλλες οι μεταφορές. Ε, πολλές φορές μπορεί οι άνθρωποι που ζουν σε κακές περιοχές να έχουν έτσι πρόσβαση σε δουλειά. Ε, άλλες φορές ε, λοιπόν είναι η βελτίωση της υποδομής. γενικά Υπάρχουν διάφορες μορφές παρέμβασης στις μικρές περιοχές. Χρειάζεται ολοκληρωμένη σκέψη, αλλά σε ψηλότερο επίπεδο. Άλλη απάντηση, παρακαλώ. Αν διαφωνήσω κατά κάποιο τρόπο ή δώσω μια άλλη διάσταση στα σχόλια. Αν δούμε την αξιολόγηση των εμπειρογνωμόνων του Urban 2 ε, βλέπουμε ότι τα διάφορα επίπεδα έχουν διάφορους, διαφορετικούς ρόλους. Τα ευρήματα έδειξαν ότι η εμπλοκή της ε, τοπικής κοινωνίας ήταν καλή σε τοπικές δράσεις αλλά όχι στην αναγέννηση της γενικότερης οικονομίας. Ε, έχει λοιπόν ε, κάποιο νόημα να αντιμετωπίσουμε οικονομικά θέματα σε ευρύτερο επίπεδο πόλης αλλά τα προβλήματα τα τοπικά να αντιμετωπίζονται σε τοπικό επίπεδο. Πολλές φορές ε, μπορεί κανείς να έχει στο μυαλό του ε, συγκεκριμένα προβλήματα στο δρόμο του, αλλά όταν του δίνουμε την ευρύτερη εικόνα να χάνεται. Εγώ μεγάλωσα στο Λονδίνο και εκεί ε, παρακολούθησα το πρόγραμμα Stockwell. Οι ντόπιοι ε, είχαν πολλές γνώσεις όταν μιλούσαν για το Stockwell αλλά όταν πήγανε στο πρόγραμμα, στην Επιτροπή για το πρόγραμμα του Λονδίνου είχαν χαθεί τελείω. Δεν είχαν ιδέα πώς ε, να αντιμετωπίσουν και να χειριστούν τα μεγαλύτερα προγράμματα για ευρύτερη περιοχή. Άρα το κάθε μέγεθος περιοχής έχει άλλο ε, πλεονέκτημα. Οι μικρές περιοχές αντιμετωπίζουν τοπικά προβλήματα, οι μεγάλες οικονομικά προβλήματα. Ευχαριστούμε. Σύντομα να πω ότι οι καινοτόμε δράσει που υποστηρίζει, στήριξε το Urban έχουν ένα συγκεκριμένο ρόλο να παίξουν. Στις πόλεις υπάρχει συγκεκριμένα μια άμεση σχέση με την Επιτροπή μέσω του Urban, η οποία πρόθεσε την καινοτομία. Και υπάρχει και μια σύνδεση μέσα από τα πλαίσια του δικτύου με άλλες πόλεις που έχουν τα ίδια προβλήματα. Ε, δεύτερον, υπάρχει μια φιλόδοξη ατζέντα στο Έρμπαν, όπως υπόθηκε. Όμως, είναι σημαντικό να μην μειωθεί η διάσταση η αστική του Έρμπαν μόνο στην ε, και τη δικτύωση. Ευχαριστούμε. Αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει το λόγο, ο κύριος Φανίστερόη έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τους ε, ομιλητές ε, που μας παρουσίασαν μια καινούργια αρχιτεκτονική. Σε αυτό που είπε ο κύριος ε, Όλτρεχτ, ε, αν διαβάσω την έκθεση συνοχής, η έμφαση δίνεται στις μεταρρυθμίσεις και το σχέδιο μεταρρύθμισης. Άρα πρέπει να υπογραφούν ε, συμβάσεις ε, και θα ήθελα να ξέρω ποιες είναι, ποια είναι η δική σας εκτίμηση γιατί έχουμε την εντύπωση εμείς ότι η εδαφική εφαρμογή, εμπλοκή των ε, περιφερειών, των διαφόρων αστικών και αγροτικών περιοχών θα πρέπει να έχει ένα ρόλο να παίξει ε, χάρη ας πούμε στην αποκέντρωση όπως έγινε για κάποιες πόλεις στις ε, αλλά πρέπει ταυτόχρονα να έχουμε μια πιο συγκεκριμένη ιδέα σχετικά με τον τύπο των ε, διαπραγματεύσεων που πρέπει να γίνουν από τη στιγμή που σταματά το σχέδιο. Υπάρχει κάποιο ας πούμε σύμφωνο εδευτικό αναχώρα. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Είναι ένα πακέτο το οποίο πρέπει να είναι ολοκληρωμένο. Και θα ήθελα να ξέρω αν προχωρούμε μέσα από το διαχωρισμό ή από την ολοκλήρωση. Ε, ευχαριστούμε. Ο κύριος Ζέλερ. Äh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όλες οι παρουσιάσεις των επιρρογνώμων έδειξαν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα αναγνώρισης. παρουσιάστηκαν όλα πολύ ρεαλιστικά και είναι ακριβώς αυτά που αντιμετωπίζουμε και, δεν, και γνωρίζουμε ξεκάθαρα στις πόλεις και το αστικά ε, κέντρα. Όμως, ε, σε όλη τη συζήτηση φαίνεται ότι υπάρχει ε, πρόβλημα εφαρμογής που από τη μία απαιτεί εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη μία πλευρά, είπαμε, για το πώς θα γίνει η εφαρμογή. Για παράδειγμα, όταν μιλάμε για στόχους ε, της ε, στρατηγικής 2020, ε, μπορεί οι αστικές περιοχές και οι κοινότητες που είναι υπεύθυνε για τέτοια σχέδια να ρωτηθούν αν γνωρίζουν τίποτα για αυτά. Θα δείτε ότι δεν ξέρουν και πολλά. Στο Βερολίνο, ας πούμε, από που είμαι εγώ, τα πράγματα είναι καλύτερα από τις άλλες πόλεις, γιατί είμαστε μια πόλη εν πόλη. Είμαστε μια πόλη κρατήδιο ε, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Και έτσι λοιπόν η περιφερειακή κυβέρνηση και οι δημοτικές ε, και αρχές ε, μπορούν να συμφωνήσουν στα προγράμματα. Στα άλλα κρατήδια είναι διαφορετικά τα πράγματα. για κάποια θέματα είναι υπεύθυνα τα κρατήδια και χρησιμοποιούν τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, π.χ. για την ανέχεια. Ε, υπάρχουν κάποια σχέδια επένδυσης ε, για το πώς θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ε, τα κονδύλια και πώς θα κατευθυνθούν στις πόλεις. Από την άλλη, επειδή οι πόλεις είναι στα πλαίσια της επικουρικότητας οι υπεύθυνες, έχουν μεν την εφαρμογή, αλλά δεν παίρνουν τόσε αρμοδιότητε σε επίπεδο επένδυση. Αυτά λοιπόν είναι κοινωνικά προβλήματα που ζητάνε οι κοινωνικά σχέδια, η εργασία με τους νέους, τα σχολεία, ε, η σωστή διατήρηση της ε, αστικής ε, υποδομής. Αυτά είναι πράγματα που χρειάζονται να χρηματοδοτούνται συνεχώς γιατί υπάρχει υποχρηματοδότηση από είναι μια χρόνια κατάσταση αυτή. Από τη δική μου πόλη συμπεραίνω ότι τουλάχιστον ε, για τις, ε, ε, για τους διάφορους δήμους ε, δεν υπάρχει αναφορά στο ευρωπαϊκό επίπεδο γιατί τα θεωρούν όλα αυτά πολύ βαρετά και δύσκολα, ότι δεν είναι βιώσιμα και έτσι όταν πάμε στην χρηματοδότηση έρχεται το μεγάλο χάσμα δεν μπορεί κανείς πλέον να εγγυηθεί ότι οι προσδοκίες που θα γεννηθούν στον τόπιο πληθυσμό τελικά θα ικανοποιηθούν θα εκπληρωθούν. Αυτό που ουσιαστικά θέλω να πω εδώ είναι ότι πρέπει να έχουμε σωστή επικοινωνία με εκείνους οι οποίοι εφαρμόζουν. Αυτό ε, πρέπει να γίνει εξ αρχής για να είναι σωστή η επικοινωνία. Πρέπει να δούμε ποιοι είναι αυτοί που ε, ουσιαστικά τρέχουν τα επιχειρησιακά προγράμματα στις περιφέρειες. Στην ε, Γερμανία δεν είναι οι πόλεις, είναι τα κρατήδια και ε, αυτοί είναι που θα θέσουν τις προτεραιότητες και δεν θα πρέπει να κατακαιρματίζεται αυτό σε πιο τοπικό επίπεδο. Έτσι λοιπόν όταν μιλάμε για τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020 για τα μελλοντικά επιχειρησιακά προγράμματα και την εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών στο σύνολό τους πρέπει πάντοτε στο προσκήνιο να έχουμε την ανάγκη να παρουσιάζονται σωστά τα πράγματα σε αυτούς που εφαρμόζουν σε κάποια φάση που θα μπορούν να αντιδράσουν σωστά. Έτσι λοιπόν ε, τίθεται το ερώτημα πώς ε, φτάνουμε εκεί όταν είμαστε στη φάση εφαρμογής και όχι στην φάση προετοιμασίας. Στη φάση προετοιμασίας είναι που πρέπει να γίνει ο διάλογος. Και να ανοίξουμε το δρόμο έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν οι πόροι όπως γίνεται, όπως πρέπει και να γίνουν τα προγράμματα όπως πρέπει και να μην λέμε στο τέλος ότι δεν είχαμε τη δυνατότητα ή τη δύναμη να κάνουμε αυτό που έπρεπε. Ευχαριστούμε τον κύριο Τσέλερ, η αντίδραση των εμπειρογνωμόνων. Πολύ σύντομα για την του κύριου Βανλίστελόε. Η πέμπτη έκθεση για τη συνοχή περίχε πρόταση η περισσότερη σύνδεση της πολιτικής συνοχής με την ατζέντα 2020 μέσω ενός κοινού στρατηγικού πλαισίου και συνεργασιών, επενδύσεων και το καθεξής. Με την έκθεση για τη συνοχή ξεκίνησε ένας δημόσιος διάλογος. Αυτά θα τα ξαναπούμε στο τέταρτο φόρουμ για τη συνοχή όπου θα συζητήσουμε τις λεπτομέρειες των εθνικών επενδυτικών συμβάσεων. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στο πλαίσιο του γενικότερου διαλόγου. Άλλωστε, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε σχόλια τα οποία δέχτηκε η Κομισιόν. Σίγουρα η εμπλοκή των τοπικών παραγόντων είναι κρίσιμη για την επιτυχία της Ατζέντας 2020. Το ερώτημα για μας είναι από εδώ και πέρα πώς όλα αυτά θα γίνουν στην πράξη βάσει των στρατηγικών κειμένων που υποβάλαμε στο πλαίσιο της πέμπτης έκθεσης. Χρειάζεται να τα συγκεκριμενοποιήσουμε όλα αυτά. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένες προτάσεις ε, βάσει και των αποτελεσμάτων του δημοσίου διαλόγου. Σύμφωνα πολύ με τον κύριο Τσέλερ υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των διαφορετικών διοικητικών επιπέδων. Δεν ξέρω πώς θα συνδυαστούν όλα αυτά. Υπάρχει ανάγκη να λάβουμε υπόψη μας τις πόλεις. Μετά οι πόλεις θα μας πούνε μετά πώς θα συγκεράσουμε τα συμφέροντά μας με αυτά των περιφερειών κλπ. Θα χαθούμε μέσα σε όλο αυτό. Πιστεύω ότι χρειάζεται θέσπιση σαφών κανόνων σε κοινοτικό επίπεδο, ώστε οι διάφορες, ε, τα διάφορα επίπεδα διακυβέρνηση να ξέρουν τι θα κάνουν μετά να εμπλακούν οι ενώσεις των ε, δήμων. Μπορούμε να βρούμε τέτοιες ρυθμίσεις για να συνεργαστούν όλοι με όλους. Και αυτό θα ήταν καλό και για τις περιφέρειες. Αν τα σχέδια αυτά δηλαδή ε, υλοποιηθούν εν τέλει. Σύμφωνα με τον κύριο Ζελέρ, η ενοποίηση τελικώς συμβαίνει σε συγκεκριμένο πάντα τόπο. Είναι λοιπόν ανάγκη προφανώς να εμπλακούν οι ερετοί τοπικοί άρχοντες και διαχειριστές ώστε να πετύχουμε συγκεκριμένα τα αποτελέσματα αυτά τα εστιασμένα αποτελέσματα που θέλουμε όπως είπε και ο κύριος Σόσιτς η λεγόμενη αιρεσιμότητα έτσι όπως τη βλέπει η Κομισιόν πόροι ε, χορηγούνται βάσει ενός ολοκληρωμένου αναπτυξικού σχεδίου σε συγκεκριμένους λειτουργικούς τομείς. Αυτό νομίζω είναι ένα δυνατό εργαλείο. ευχαριστώ. Άλλος. Ένα γενικό σχόλιο παρατηρώντας τις ε, εξελίξεις στο αστικό τοπίο στη χώρα μου τα τελευταία χρόνια πρέπει να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της εκπαίδευσης, της ε, κατάρτισης, της ομάδας έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Βοήθησε επίσης του ανθρώπους να εστιάσουν την προσοχή τους σε συγκεκριμένους στόχους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε ακριβώ το πλαίσιο με στο οποίο εμείς αναλάβαμε δράσεις. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία σε πολλαπλά επίπεδα από τη γειτονιά στην πόλη και πιο ψηλά να υπάρχει από εδώ και πέρα για άλλη μια φορά ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Πρώτος, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τους εμπειρογνώμονες για τη συμβολή τους. Θα ήθελα να χαιρετήσω εδώ δύο Αυστριακούς δημαρχούς, οι οποίοι κέρδισαν το βραβείο Δήμαρχος της Χρονιάς 2011 11 της Επιτροπής των Περιφερειών. Συνεχίζουμε. Επόμενο σημείο στη μέση διάταξη. Σημείο 19. Ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Ρούντελφ Νίσλερ, Διευθυντή Συντονισμού Πολιτικής της Γενικής Διευθύνσης Ρέτζιο, σχετικά με την ε, ανταπόκριση σε πολιτικό επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την συνοχή στην οικονομική κρίση. Κύριε Νίσλε, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τα επόμενα λεπτά θα σας παρουσιάσω την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την συμβολή της περιφερειακής πολιτικής στην προσπάθεια των κρατών μελών να προκρίνουν μέτρα για να αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2009. Όπως όλοι γνωρίζετε, η, πολιτική συνοχής υλοποιήθηκε για να αντιμετωπιστεί η κρίση. Η κεντρική ιδέα τότε ήταν να κινητοποιήσουμε μέρος των διαθέσιμων πόρων στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, καθώς και άλλα υποστηρικτικά μέτρα, τα οποία ε, θα μπορούσαν καλύτερα να προσαρμόσουν τα κρατημέλη στις ανάγκες. Τώρα το πλαίσιο αποσαφηνίστηκε από νωρίς λόγω της κρίσης. Διαπιστώσαμε τα προβλήματα των τραπεζών που έκλεισαν τις στρόφιγγες του δανεισμού. Παρατηρήσαμε επίσης ότι σε επίπεδο κράτους μέλους οι περιφέρειες αντιμετώπισαν παρόμοια προβλήματα με αποτέλεσμα στο πλαίσιο της ε, πολιτικής συνοχής ε, οι δυνατότητες χρηματοδότησης να είναι ακόμη λιγότερες και να κινδυνεύουν συγκεκριμένα προγράμματα. Ο στόχος της πολιτικής συνοχής ήταν να συνδράμει δεδομένη της κατάστασης χωρίς να υπορμευθούν, ε, να διοικηθούν οι μακροπρόθεσμοι στόχοι. Ο στόχος της πολιτικής ε, συνοχής είναι να επιταχυνθούν οι διαδικασίες μέσω απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών οι επικεφαλής των προγραμμάτων να κινηθούν με μεγαλύτερη ευελιξία συναρτήσει των ε, αναγκών και των περιοχών που επηρεάστηκαν από την κρίση να εξασφαλιστεί υπαρκής χρηματοδότηση από τα πρώτα στάδια και να δημιουργηθούν νέες επιλέξιμες ενέργειες στο τομέα της ε, ενεργειακής απόδοσης καθώς και στην εξασφάλιση τεχνικής υποστήριξης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γενικώ 13 επιμέρους μέτρα προτάθηκαν πλέον στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής ε, και συγκεκριμένα στο πλαίσιο της πολιτικής αντιμετώπισης της κρίσης. ...6,25 δισεκατομμύρια ευρώ προκλήθηκαν υπέρ του περιφερικού και του Κοινωνικού Ταμείου για να χρηματοδοτηθούν, για να χρηματοδοτηθούν τα σχετικά προγράμματα. Συνολικά, ο προπολογισμό έφτασε στα 11 δισεκατομμύρια ευρώ. Όπω ξέρετε, οι προκαταβολέ είναι πολύ σημαντικέ. Είναι μια κυλιόμενη χρηματοδοτική μέθοδο. Τώρα έγιναν και 7 άλλε αλλαγέ στον δρόμο τη απλούστευση των διαδικασιών για να προσδώσουμε μεγαλύτερη ευελιξία στην χορήγηση παράδειγμα των κοινωτικών ενισχύσεων πετράπη, δηλαδή η καταβολή προκαταβολών σε μεγάλα επενδυτικά σχέδια ε, στο πλαίσιο των προγραμμάτων ενεργειακής απόδοσης και εξοικονομής ενέργειας. Τα κονδύλια για την ε, τεχνική βοήθεια και αυτά βοήθησαν να επιταχυνθούν προγράμματα μέσω του Jaspers που χρηματοδοτεί και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και επίσης εξασφαλίσαμε και ε, ενίσχυση από το Τζέρμι και από το Τζέσικα. Στο πρόγραμμα ανάκαμψη η πολιτική συνοχή κατέδειξε ότι είναι αρκετά ευέλικτη και ότι προσαρμόζεται για να επιτύχει και βραχυπρόθεσμου στόχους. Η επιτυχία αυτή στον τομέα της ευελιξία και της ταχύτητας εξασφαλίστηκε χάρη και την ποιότητα τη δουλειά που έγινε μεταξύ των θεσμικών οργάνων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, την επικοδομητική συνεργασία δηλαδή που είχαμε εμεί ω θεσμικοί εταίροι, το Συμβούλιο συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή των Περιφερειών και η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Ανταποκριθήκαμε λοιπόν γρήγορα και νομίζω με το σωστό τρόπο. Η ευελιξία λοιπόν κατέστη δυνατή ακριβώς επειδή όλοι εργαστήκαμε προς την ίδια κατεύθυνση. Με την παρούσα έκθεση σας παρουσιάζουμε αυτό το οποίο έπρεξε η Κομισιόν ανταποκρινόμενη και σε έκκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης του, του πακέτου. Είχε ζητήσει δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υποβληθεί σχετική έκθεση το φθινόπωρο του 2010 και αυτό ακριβώς κάνουμε αυτή τη στιγμή. Οι πηγές των δεδομένων για την έκθεση. Αντλήθηκαν από τα στοιχεία που έδωσαν τα κρατημέλη για την στρατηγική έκθεση. Όπως γνωρίζετε, η στρατηγική έκθεση ε, βασίστηκε σε 27 εθνικές συνεισφορές και ζητήσαμε από τα κράτη-μέλη το καθένα σε ένα, στο δικό του κεφάλαιο να μας παρουσιάσει τα μέτρα και το πώ χρησιμοποιούν τα διαρθρωτικά ταμεία για να αντιμετωπίσουν την κρίση. Επιτρέψτε μου λοιπόν να πω δύο λόγια για τα βασικά μέτρα, για του βασικού τομεί και να δώσω και μερικά παραδείγματα για τα όσα έκαναν τα κράτη-μέλη χάρη στην ενίσχυση που του παρέσχομαι. Για παράδειγμα, στον τομέα των προκαταβολών, τα 6,2 δισεκατομμύρια ε, που σας προανέφερα που καταβάλαμε τον Ιούνιο του 2009 ακριβώς για να καλύψουμε τι ανάγκε χρηματοδότηση προχρηματοδότηση και να επιταχύνουμε την υλοποίηση. Γενικά είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την χρησιμοποίηση αυτή τη επιπλέον χρηματοδότηση. Γιατί έτσι προλάβαμε και την απώλεια κονδυλίων λόγω του κανόνα νη συν Το λέω αυτό διότι θα ήταν εξαιρετικά τυχής ε, εξέλιξη εν μέσω της κρίσης να χαθούν ακριβώς κονδύλια από τα κράτη-μέλη λόγω του κανόνα νη συν και μόνο. Έτσι λοιπόν βγήκαν από αυτή την ε, δύσκολη θέση ορισμένα κράτη-μέλη και αυτό το λέει και η έκθεση. Τα κράτη-μέλη χρησιμοποίησαν τα κονδύλια αυτά κυρίως σε έργα όπου έλειπαν ακόμη πιο έντονα οι εθνικοί πόροι σε τοπικό επίπεδο, τοπική αυτοδιοίκηση, οι μη κυβερνητικέ οργανώσει, για παράδειγμα έκαναν αυτό. Οι προκαταβολές επίσης χρησιμοποιήθηκαν για να υποστηριχθούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να ενισχύσουν επίσης εθνικά προγράμματα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στην Πολωνία και την Ιστορία, για παράδειγμα, τα σχετικά εθνικά προγράμματα αναπροσαρμόστηκαν για να επικεντρωθούν στις πιο ευάλωτες ομάδες επιχειρήσεων μεταξύ αυτών και μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να περιοριστούν ακριβώς οι επιπτώσεις της κρίσης σε αυτές τις ομάδες επιχειρήσεων. Τα κράτη-μέλη θεωρούν ότι υπήρξαν θετικά αποτελέσματα. Επίσης στον τομέα της ρευστότητα και στην υποστήριξη επενδύσεων. Για παράδειγμα, στην Ιταλία είχαμε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα για την έρευνα και την ανταγωνιστικότητα. Στην Ελλάδα οι προκαταβολές επέτρεψαν την καταβολή ενισχύσεων σε δικαιούχους σε τρεις τομείς προτεραιότητας. Προγράμματα προμηθειών, προγράμματα υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω επαγγελματική κατάρτιση και ούτω καθεξής. Τώρα στον δεύτερο τομέα, προσαρμογή των προτεραιοτήτων των επιχειρησιακών προγραμμάτων και δυνατότητα επαναπρογραμματισμού, τροποποίηση του προγραμματισμού. Η Κομισιόν είχε συστήσει για την αντιμετώπιση της κρίσης να δούμε με ευελιξία μερικά θέματα και να ικανοποιήσουμε ταχύτατα ε, δύο αιτήματα από κράτη-μέλη που θέλουν να επαναπροσανατολίσουν, να επαναδημορφώσουν τα επιχειρησιακά τους προγράμματα. Επιβεβαιώσαμε ομοφόνος τους στόχους των εθνικών στρατηγικών πλαισίων. Όλοι υποστηρίξαμε ότι οι βασικές προτεραιότητες πρέπει να παραμείνουν ως έχουν βάσει του στόχου της Λισαβόνας της ε, δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Λοιπόν, γενικά σε στρατηγικό επίπεδο είπαμε ότι δεν θα τροποποιήσουμε τους στόχους μας, ότι πρέπει να μείνουμε προσυλλομένοι στους στόχους των διευθυντικών ταμείων. Παρ' αυτά, τα κράτη-μέλη έκαναν μερικές στοχευμένες αναδομής των επιχειρησιακών τους προγραμμάτων και όταν λέω άλλαξαν ε, προγράμματα δεν άλλαξαν όλα τα προγράμματα βεβαίω. έγιναν κάποιες τροποποιήσεις σε 17 μέλη, κάτι μέλη τα οποία αποτελούν ακριβώς ε, την απάντηση αυτών των κρατών μελών στην κρίση Αυτές οι εσωτερικές αναπροσαρμογές ανιστικούν σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Παράδειγμα, στο, στην υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για να προληφθεί η απώλεια θέσεων εργασίας. Αυτό ήταν ένα μέτρο προτεραιότητας. Επίσης δεχθήκαμε να είναι επιλέξιμες ε, πρωτοβουλίε στον τομέα της οικονομής ενέργειας στο, στις κατοικίες. Επίσης, εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την ευελιξία που έδειξαν τα κατημέλη και για την ταχύτητα με την οποία η Κομισιόν ε, ενέκρινε τα μέτρα αυτά. Τα μέτρα για την ενεργειακή απόδοση, για παράδειγμα, ε, με να σχολιάσω λίγο περισσότερο το θέμα γιατί νομίζω ότι είναι εξαιρετικά επίκαιρο και ενδιαφέρον. Όπως γνωρίζετε ο σχετικός κανονισμός τροποποιήθηκε ώστε οι ανανόσιμες μορφές ενέργειας και η ενεργειακή απόδοση να ενταχθούν στα προγράμματα βελτίωσης των κατοικιών με προπολογισμό 4% του συνολικού προπολογισμού. θεωρητικά αυτό θα μπορούσε να φτάσει στα 8 δις ευρώ. Τα νέα κριτήρια επιλεξιμότητας εισήχθησαν όπως ε, γνωρίζετε στο πλαίσιο του πακέτου για την αντιμετώπιση της κρίσης συγκεκριμένα όπως προείπα και για να ενισχυθεί και η στρατηγική για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος. Είναι καλό έστω και εν μέσω κρίσης να θυμίζει κανείς ότι υπάρχει ένας στρατηγικός προσανατολισμός, ένας στρατηγικός στόχος ο οποίος πρέπει να συνεχίσει να μας απασχολεί και μακροπρόθεσμα. Επίσης, εγκρίναμε και άλλα συγκεκριμένα μέτρα. Για παράδειγμα, υποστήριξη της βιομηχανίας, της οποίας ο ρόλος είναι γνωστός στην δημιουργία θέσεων εργασία αλλά και στο περιβάλλον. Υποστηρίξαμε την βραχυπρόθεσμη δημιουργία θέσεων εργασία. Με τα μέτρα μέσω μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο. Ας πούμε, αντλίες θερμότητας ή ηλιακά πάνελ σε κατοικίες. Αυτό δίνει δουλειά πολύ συχνά σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες ακριβώς δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Επίσης πιστεύουμε ότι αυτές οι επενδύσεις αν διαδοθούν, θα έχουν και ουσιαστική συνεισφορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και έτσι ενδέχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναδειχθεί σε ηγέτη, σε πρωτοπόρο σε αυτόν τον τομέα, στη συγκεκριμένη τεχνολογία δηλαδή της ενεργειακής απόδοσης. Για να ενισχύσουμε περαιτέρω αυτές τις δράσεις σε επακολουθή δράση επιτρέψαμε τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης να είναι επίσης επιλέξιμα για χρηματοδότηση από τα διάφορα χρηματοδοτικά μέσα με συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων η οποία μας βοήθησε πολύ στην δρομολόγηση αυτών των μέτρων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Τζέσικα συγκεκριμένα όπως ε, προείπα αλλά και για τα νέα χρηματοδοτικά μέτρα, το financial engineering που προβλέπει ο κρονισμό. 14 κρατημέλη προκειμένου ανέφεραν ότι αξιοποίησαν αμέσως αυτές τις ευκαιρίες επενδύσεων δηλαδή στην ενεργειακή απόδοση και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο τομέα αυτό ξεκινήσαμε ουσιαστικά από το μηδέν. Τα μέτρα λοιπόν αυτά θα απαιτήσουν κάποιο χρόνο μέχρι να εξαπλωθούν και να γίνουν αισθητά. Αυτό λοιπόν ήταν ένα θετικό μέτρο. Επιπλέον, προσπαθήσαμε επίσης να υποβοηθήσουμε τους εναλλακτικού τρόπου χρηματοδότηση. Μαζί με την ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προσπαθήσαμε να προωθήσουμε το Jeremy, να ενισχύσουμε δηλαδή τι μικρομεσαίε επιχειρήσει και στο πλαίσιο αυτό εξασφαλίζουμε πλέον τεχνική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προχωρήσει το μέτρο. 12 κρατη εδώ αξιοποίησαν τις δυνατότητες και χρησιμοποίησαν τις πρωτοβουλίες του Τζέρεμι ακριβώς για να υποστηρίξουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το Τζέσικα επίσης επιταχύνθηκε θεματικά θα έλεγα. Όπως ξέρετε το Τζέσικα ήταν πρωτοβουλία που προστάθηκε καθυστερημένα στον κανονισμό. Ξεκίνησε με σχετικά αργά, όμως προς έκπληξή μας και ίσως και χάρη στην κρίση τα αποτελέσματα είναι πολύ καλά. Έχουμε αυτή τη στιγμή 21 μέτρα που χρηματοδοτήθηκαν από το ε, Τζέσικα. Τα νέα μάλιστα τα διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στα αντίστοιχα κράτη-μέλη. Τέλος, την τεχνική βοήθεια. Βελτιώσαμε τις δυνατότητές μας στο πλαίσιο της πρωτοβουλία Jasper και πάλι με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αλλά και με άλλους ε, εταίρους. Την ε, EBRD και το KFW, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης. Ήδη 85 πυρογνώμονες δουλεύουν για μας οι οποίοι υποστηρίζουν την προετοιμασία των προγραμμάτων στην Ευρώπη των 12 και προσπαθούν επίσης να επιταχύνουν την υλοποίηση των μεγαλύτερων προγραμμάτων και φροντίζουν και για την ποιότητα. Αυτά είναι τα βασικά μέτρα του πρώτου γύρου των μέτρων για την ανάκαμψη από την κρίση μετά από αυτά όμως, όπως γνωρίζετε, τροποποιήθηκε πάλι ο κανονισμός για τους σκοπούς ε, της απλούστευσης. Ήταν, ήταν το περίφημο πακέτο απλούστευσης που αρχίζει να ισχύει από φέτος. Και εδώ σκοπεύουμε να ενισχύσουμε χώρες που αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις της κρίσης. Τα μέτρα αυτά εδώ όμως είναι μικρότερης κλίμακας και αποσκοπούν ειδικότερα στην Λετωνία, στην ε, Ρουμανία, την Πολωνία ε, πέντε χώρες ε, συνολικά και για 370 εκατομμύρια ευρώ συμπληρωματική προκαταβολή. Και τούτο διότι αυτές οι πέντε χώρε συγκεκριμένα είναι οι χώρες που επλήγησαν περισσότερο από κάθε άλλη, ειδικά στον τομέα της απασχόλησης. Ειδικά για την Ελλάδα, όπω γνωρίζετε, υπάρχει το γνωστό μνημόνιο το οποίο συνομολογήθηκε το Μέο του 2010 και το οποίο καθορίζει τους στόχους του οικονομικού προγράμματος της κυβέρνησης και το οποίο υποστηρίζεται από την ε, ομάδα των ευρωπαϊκών κρατών μέσω μια ε, συμφωνία δανειακή διευκόλυνση. Το μνημόνιο προβλέπει συγκεκριμένε δράσει ε, των διαρθρωτικών ταμείων. Πολύ σημαντικέ είναι η δημιουργία μια ειδική ομάδα έργου η οποία λειτουργεί και αναφέρεται κατευθείαν στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Εκεί υπάρχει προσωπικό της Κομισιόν το οποίο βοηθάει στην προετοιμασία, την κατάρτιση ε, των αποφάσεων που αφορούν την πολιτική συνοχή. Και αυτό το μέτρο θα επιταχύνει πιστεύω την υλοποίηση, μάλλον την προετοιμασία και την υλοποίηση των προγραμμάτων στην Ελλάδα χάρη στα ταμεία χαρτοφυλακή όπω τα λέμε, τα οποία χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία και τα οποία επενδύουν μέσω συγκεκριμένων χρηματοδοτικών μηχανισμών σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα της αστικής ή της ενεργειακής απόδοσης. Αυτό σας δίνει, πιστεύω, μια συνολική εικόνα του τι κάνει η πολιτική συνοχής για να υποστηρίξει τα κράτη-μέλη αλλά και τις περιφέρειες στον αγώνα που κάνουν για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της κρίσης. Τα κράτη-μέλη μας λένε ότι είναι πολύ ικανοποιημένα από την ταχύτητα της απάντησής μας όσο και από την ευελιξία. Εμείς αυτό κάνουμε. Προτείναμε να βρει φάσμα λύσεων, προτάσεων. Ξέραμε ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν όλοι όλες τις δυνατότητες, αλλά τουλάχιστον τα κράτη-μέλη είχαν την δυνατότητα να επιλέξουν τους τομείς στους οποίους θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν κάποια κονδύλια. Και αυτό είχε πολύ θετικές επιπτώσεις. Το πρόγραμμα λοιπόν για την αντιμετώπιση της κρίσης πήγε καλά. Θα έλεγα λοιπόν ότι Εν γέννη, αν θέλαμε να απαντήσουμε στο γενικό ερώτημα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η πολιτική συνοχή, που είναι μια μακροπρόθεσμη πολιτική, με μακροπρόθεσμου στόχου. Αν μπορεί λοιπόν η πολιτική αυτή να συνδράμει και στην βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση μια ε, παροδική βεβαίω κρίση, τότε η απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα ήταν ναι. Σίγουρα λοιπόν η πολιτική συνοχή συνέβαλε θετικότητα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Μανέσκου καταρχήν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Νίσλερ για την παρουσίασή του. Διάβασα τον γράφο εργασία που κατάρτισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από όσο κατάλαβα η υποβολή εκθέσεων από τα κράτη-μέλη ήταν κατακαιρματισμένη και γι' αυτό η Κομισιόν είχε δυσκολία στο να ποσοτικοποιήσει τον αντίκτυπο των μέτρων που έλαβαν τα κράτη-μέλη για την καταπολέμηση της κρίσης τα τελευταία τρία έτη. Στο πλαίσιο αυτό και ε, ιδίω τα πέντε κράτη-μέλη που χτυπήθηκαν ιδιαίτερα από την κρίση έλαβαν σημαντική ε, οικονομική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω, θα ήταν δίκαιο για αυτά τα κράτη-μέλη να αναφέρουν ποια μέτρα έλαβαν ε, για να δούμε αν έλαβαν τα σωστά μέσα και αν χρησιμοποίησαν ε, ορθά τα χρήματα για τους σκοπούς που είχαν καθοριστεί. Η πρώτη μου ερώτηση είναι γιατί πιστεύετε ότι η Κομισιόν είναι σε θέση να δώσει μία πλήρη και ολοκληρωτική αξιολόγηση στο Κοινοβούλιο. Εδώ, το έγγραφο αυτό προκύπτει από πληροφορίες ε, των κρατών μελών μέσω των Εθνικών Στρατηγικών Προγραμμάτων του 2009. Έχουμε υποβολή εκθέσεων για, τα, ε, για τους πόρους που δόθηκαν ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, για τα μέτρα που υλοποιήθηκαν για την οικονομική ανάπτυξη. Από ό,τι κατάλαβα, τα στοιχεία της Ρουμανίας, Λουχάρη, δεν συνδέονται πάντα με την οικονομική πραγματικότητα. Θα ήθελα να μου πει η Κομισιόν, αν κατά κατάρτιση αυτών των εκθέσεων περιορίστηκε η Κομισιόν στις πληροφορίες που έλαβε από τα κράτη-μέλη και μόνο δηλαδή πληροφορίες που ενίοτε μπορεί να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ή εάν Κομισιόν έχετε κάποιες πληροφορίες ή κάποια σημάδια ότι υπάρχουν λάθη στα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά την εφαρμογή την απορρόφηση και στην περίπτωση αυτή η Κομισιόν θα εξετάσει στενότερα τι συμβαίνει σε αυτά τα κράτη-μέλη. Θα παρακολουθήσει η ίδια αυτά τα ή η Κομισιόν απλώ ε, περιορίζεται σε αυτέ τι πληροφορίε που λαμβάνει από τα συγκεκριμένα κράτη-μέλη. Και κατόπιν έχουμε ένα φαυλοκύκλο. Παραπονιόμαστε ότι τα κράτη-μέλη δεν ε, υποβάλλουν τι ε, σωστέ εκθέσει. αλλά δεν κάνουμε τίποτα για να διορθώσουμε την κατάσταση. Έτσι λοιπόν, έρχομαι στη δεύτερη ερώτηση. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η Κομισιόν θα πρέπει να εμπλέκεται περισσότερο στην παρακολούθηση της κατάστασης. Ευχαριστώ. Κυρία Σρέντερ, ευχαριστώ. Θεωρώ ότι η προηγούμενη μιλήτρια έθεσε μια πολύ καλή ερώτηση και εγώ να συμπληρώσω κάτι. Πρώτον, μάλλον ε, ο εισηγητής έδειξε τις θετικές και όχι τις αρνητικές πλευρές αυτού που έγινε. Και αυτά θα πρέπει να τα κοιτάξουμε πιο συγκεκριμένα. Συγκεκριμένα στη συγχρηματοδότηση για τα κράτη-μέλη ε, δεν ε, χρησιμοποιήθηκαν όλες τις ε, δυνατότητες. Είτε δεν δόθηκαν χρήματα, είτε οι αρχές θεώρησαν ότι δεν ήταν ας πούμε ελκυστικά ε, τα κονδύλια. Το Λουξεμβούργο, πούμε, αντέδρασε, τα άλλα κράτη όχι. Ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο είχε να κάνει με τη συγκεκριμένη οικονομική συγκυρία. Ε, ας πούμε, είχε να κάνει με την ε, μηχανή των θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο, τα κτίρια κτλ. όταν έχουμε μόνο 12 κράτη-μέλη, δηλαδή το λιγότερο από τα μισά που χρησιμοποίησαν αυτό το, αυτή τη δυνατότητα, έχουμε κατανοούμε ότι είναι πολύ λίγος ο αριθμός. Γιατί δεν ε, χρησιμοποιήθηκαν, ποια ήταν η, σχέση της Κομισιόν, ποια ήταν οι επιπτώσεις... Ε? Ήταν μια ένεση ε, για την οικονομική συγκυρία. Τι ακριβώς. Κάτι άλλο που παρουσιάστηκε πολύ καλά ήταν η συνεργασία της Ευρωπαϊκής ε, Τράπεζας Επενδύσεων και του Τζάσπερς. Πόσο διαφανής ήταν αυτή η συνεργασία. Πώς, ε, ποιοι συμμετείχαν. Και η εργασία ε, επικεντρώθηκε στα απαραίτητα μέτρα για τα μεγάλα project όπου δόθηκαν πολλά ε, χρήματα και αν ε, έγινε κάτι τέτοιο έγινε σωστά επειδή ε, στις, στο περιβάλλον όταν είναι προβληματικό δεν έχουμε μια καλή εικόνα προς τα έξω υπάρχουν κάποιες θέσεις σε αυτό. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Έχουμε δύο ακόμα συνάδελφους που έχουν στο λόγο. Αν μπορούμε τώρα να κλείσουμε τον κατάλογο των ομιλητών, να ακούσουμε τους επόμενους δύο συναδέλφους, ο κύριος Φανιστερός και μετά ο κύριος Αγκουράκης. Ευχαριστώ. Εγώ έχω μια θετική αντίδραση απέναντι στην έκθεση και τις πληροφορίες ε, που δόθηκαν. Ουσιαστικά Δράξαμε από τα μαλλιά την ευκαιρία της κρίσης ε, για να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Το Συμβούλιο ήταν διστακτικό και νομίζω όμως ότι η κρίση τελικά είχε και κάποια θετικά στοιχεία. Μια άλλη θετική πτυχή 12 χώρες ε, μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν τη δυνατότητα καλύτερης ενεργειακής αποδοτικότητας. Αυτό είναι ένα καλό σημάδι για να πούμε ότι υπάρχει ε, συνεργασία μεταξύ κρατών και κομισιών για την επίτευξη των στόχων. Μιλάμε εδώ για εκθέσεις που αφορούν την εκτέλεση των ε, σχεδίων δράσεις γιατί τα κράτη-μέλη ήταν ελεύθερα να διαλέξουν από μια τεράστια γκάμα μέτρων προκειμένου να λάβουν κάποιες επιχορηγήσεις. Και 12 κράτη προχώρησαν και εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία. Έτσι λοιπόν αυτό μας οδηγεί στο να ζητήσουμε την αιρεσιμότητα. Κοιτάξτε εδώ. Θέλω να στραφώ στην Προεδρία. Μια προσωρινή επιτροπή του Κοινοβουλίου είχε ε, διοριστεί για να συζητήσει τα θέματα της κρίσης. Ε, όμως, τι γίνεται σήμερα. Ε, δηλαδή, έχουμε καλυφθεί από τις εκθέσεις, περιμένουμε να περάσει κρίση. τι εμείς τι θα γίνει με αυτή την έκθεση, θα τη λάβουμε και πότε θα φτάσει σε εμά. Σας ευχαριστώ κύριο Σογκουράκης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, ασφαλώς τα στοιχεία που μας παρουσιάστηκαν είναι σημαντικά, ε, ανταποκρίνονται προφανώς σε μια κατάσταση. Ωστόσο κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι ε, και τα μέτρα που πάρθηκαν αλλά και η έκθεση του κυρίου εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κομισιόν, δεν απαντάνε στο βασικό ερώτημα τι γίνεται με την κρίση. Και αυτό ούτε τα μέτρα βεβαίως έχουν αντιμετωπίσει την κρίση, απλώς έχουν ε, κάνει λιγότερα αισθητέ τις επιπτώσεις της κρίσης, αλλά η κρίση όπως γνωρίζετε σε όλες τις χώρες μας δυστυχώς πρέπει να πω βαθαίνει και οξύνεται ακόμα περισσότερο και φυσικά ε, ασφαλώς πάθηκαν κάποια μέτρα ας πούμε, αν ο κύριος ε, εκπρόσωπος της Κομισιόν δεν μιλούσε για την Ελλάδα, δεν θα να καν το λόγο. Έκανε λόγο για ορισμένα προγράμματα που βοήθησαν μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η βοήθεια πρέπει να ξέρετε είναι ελάχιστες, είναι ελάχιστη. Πάρα πολύ, ένας μεγάλος αριθμός από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν είναι καν σε θέση να πάρουν αυτά τα προγράμματα γιατί τα χρέη τους είναι τεράστια. Τα χρέη αυτά δεν αντιμετωπίζονται και πρέπει να, γενικά να σας πω κυρία Πρόεδρε ότι τα χρήματα για τα οποία μιλάμε, τα 327 δισεκατομμύρια, ασφαλώς είχαν σχεδιαστεί και τα προγράμματα πριν την κρίση και τα εργαλεία για τα οποία μιλάμε και τα μέτρα ενεργειακής ε, υποστήριξης είναι μέτρα που προϋπήρχαν της κρίσης, γι' αυτό και όλα η εφαρμογή, η επιτάχυνσή τους δεν πρόκειται να μας οδηγήσουν ε, έξω από την κρίση. Αυτή είναι μια πραγματικότητα και αυτό πρέπει να πάρθει υπόψη χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι εγώ προσωπικά είμαι αντίθετος ε, στα συγκεκριμένα μέτρα. Πρέπει όμως να ξέρετε ότι ε, μέτρα όπως αφορούν αυτά την απασχόληση συνδέονται με πολύ άσχημες συνθήκες εργασίας, με ευέλικτες ε, συνθήκες εργασίας και γενικά όταν έχω μια, είμαστε σε μια χώρα όπου η ανεργία έχει αυξηθεί κατά το 50% αυτά τα πράγματα είναι ελάχιστα. Άρα το ερώτημα που, για μένα, τίθεται για μένα για άλλη μια φορά είναι πώς μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει τις αιτίες της κρίσης και όχι απλώς με ορισμένα μέτρα που είναι πραγματικά, κατά τη γνώμη μου, ψίχουλα και δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα στη βάση του. Ευχαριστώ πολύ. Uh, uh, Ευχαριστώ πολύ. Θα σχολιάσει τώρα ο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όσα ακούστηκαν. Προσπαθήσω να απαντήσω στι ερωτήσει ε, του κ. Αγκουράκη και τη κ. Μανέσκου, ίσω εδώ, σε αυτή την έκθεση. Κατά κάποιο τρόπο έχετε μία ελληνική απάντηση που έχουμε από τα κράτη-μέλη για το τι έκαναν στην πραγματικότητα με την προσφορά που προήλθε από την πολιτική συνοχής για να του παρέχει υποστήριξη για τα προβλήματα που αντιμετώπισαν κατά το ξέσπασμα τη κρίση. Είναι αυτονόητο ότι φυσικά δεν έχει τελειώσει ε, όλη αυτή η ιστορία και το γνωρίζουμε ακόμη και αν ε, έχουμε προβλέψεις ε, για οικονομική ανάκαμψη και ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι ε, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες για να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουμε στην παρούσα συνθήκη σε ό,τι αφορά την υποβολή εκθέσεων. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να πούμε ότι αυτή είναι μία πρώτη έκθεση για το τι άμεσα χρησιμοποίησαν τα κράτη-μέλη από αυτή την προσφορά της πολιτικής συνοχής. Στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής έχουμε ένα σύστημα υποβολής εκθέσεων που βασίζεται σε τήσεις εκθέσεις ε, που μας στέλνονται και που μας αναφέρουν ε, ποια είναι η συνολική πρόοδος ε, στην εφαρμογή των μέτρων. Παρ' όλα αυτά θα τολμούσα να πω το εξή ότι δεν έχουμε πλέον μια διαφοροποίηση μεταξύ των συγκεκριμένων ε, μέτρων που σχετίζονται με την κρίση και μεταξύ και με αυτών που ε, των πτυχών που έχουν να κάνουν με την εφαρμογή των μέτρων. Έτσι λοιπόν ε, θεωρώ τώρα ότι ε, παρακολουθούμε και προσδίδουμε συνέχεια και σε προβλήματα και ερωτήσεις που μπορεί να ανακύψουν στα κράτη-μέλη επειδή συνεχίζονται τα προβλήματα στην πραγματική τους οικονομία. Και η πολιτική συνοχή θα αναλύσει προσεκτικά την κατάσταση και στα πλαίσια των δυνατοτήτων των μέσων που έχουμε θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε. Αλλά αυτός είναι ο κανονικός τρόπος ε, που ε, λειτουργεί η πολιτική συνοχή. Είναι δύσκολο λοιπόν ε, να διαφοροποιήσουμε περαιτέρω ζητήματα που άπτονται αποκλειστικά της κρίσης. Τώρα, τι είπε η κυρία Σρέτερ σε σχέση με τα πιο θεμελιώδη προβλήματα που είχαμε σε ορισμένα κράτη-μέλη. Παραδείγματο χάρη στο να εξεύρουμε συγχρηματοδότηση. Αλήθεια είναι. Είχαμε συναντήσει τέτοια προβλήματα, κυρίως σε ορισμένα νέα κράτη-μέλη και όπως γνωρίζετε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, ε, δημιούργησε ένα μοντέλο σημαντικής στήριξης ε, για να διασφαλίσει ότι μέτρα που χρηματοδοτούνται μέσω της πολιτικής συνοχής μπορούν να προχωρήσουν και δεν καθυστερούν λόγω της έλλειψης πολιτικής συνοχής. Έχουμε ανοιχτές πιστοτικές γραμμές για αρκετές χώρες υπό, από τις 12 χώρες και έτσι είναι δυνατό να συνεχιστεί η εφαρμογή των προγραμμάτων. Αυτό σε έναν βαθμό σχετίζεται με την κρίση. Και παρακολουθούμε την κατάσταση μαζί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πολύ προσεκτικά, προκειμένου να δούμε αν ε, εκεί εμπεριέχονται περαιτέρω κίνδυνοι σε ό,τι αφορά τώρα την ενεργειακή αποδοτικότητα. Είδαμε μια ιδιαίτερη επιλακτική επικαιροποίηση των μέτρων αυτών. Για όσο είπε ο κύριο Φανίσταλ Ταλρόη. Κατά κάποιο τρόπο ορθή είναι αυτή η κρίση. Αν δείτε τα παλιά κρατημέλη, τα 15 κρατημέλη, σε Κάποια κράτη-μέλη υπήρχαν ήδη αναπτυγμένε ε, πολιτικέ που υποστήριζαν τα μέτρα ενεργειακή αποδοτικότητα στην Γερμανία στην Αυστρία. Υπήρχαν ήδη ε, συστήματα στήριξη στι κατοχώρε. Τέτοια συστήματα που λειτουργούσαν μέσω συνδυασμού επιδοτήσεων και δανείων με ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο. Ήταν λοιπόν σαφές από την αρχή ότι οι Γερμανοί, οι Αυστριακοί δεν θα αναθετούσαν αυτό το μέτρο. Διαφορετική ήταν η κατάσταση με τη Γαλλία λόγου χάρη. Η Γαλλία χρησιμοποίησε αυτή την ευκαιρία αμέσως όταν ε, υπήρξε αυτό το άνοιγμα στον κανονισμό και τώρα σε πολλά επιχειρησιακά προγράμματα άρχισαν να αναπτύσσει μέτρα για την υποστήριξη της ε, κοινωνικής στέγασης ε, με νέες βελτιωμένες μεθόδους συνεργειακής αποδοτικότητας. Η στήριξη του πληθυσμού είναι από τα πλέον αποτελεσματικά μέτρα Αποκλείστηκαν οι οικογένειε ε, που υπέφεραν ε, από την απειλή τη στόχιας, όμω ξέρουμε από τις γαλλικές αρχές ότι σκοπεύουν ε, να παρουσιάσουν και κάποια συστήματα στήριξη που θα περιλαμβάνουν χρήματοδοτικού μηχανισμού. Αυτά τα μέτρα ενεργειακή αποδοτικότητα επίσης Ε, υιοθετήθηκαν και σε ορισμένα νέα κράτη-μέλη σε μεγαλύτερο βαθμό. Θα θυμάστε ότι υπήρχε μία διάταξη στον κανονισμό ήδη, η οποία επέτρεπε σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις ε, τα, να ενεργοποιηθούν τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στα κράτη-μέλη και για την επένδυση σε ενεργειακή αποδοτικότητα στα πλαίσια της αναγέννησης των πόλεων. Αυτό το είδαμε τώρα με το άνοιγμα του κανονισμού ότι πιο σημαντικά μέτρα εφαρμόστηκαν στα κράτη-μέλη. Και φυσικά υπήρξε και συγχρηματοδότηση και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και σε ορισμένε περιπτώσει συμμετέχουν και εθνικέ τράπεζε. Και βλέπουμε ότι αυτά τα μέτρα κερδίζουν έδαφος τους επόμενου μήνες. Για να κρίνουμε τα μέτρα αυτολογικά. Στο στάδιο αυτό δεν πρέπει να προβούμε σε συγκρίσεις της αποτελεσματικής υιοθέτηση με ε, τις δαπάνες και το υποθετικό νούμερο των 6 δισεκατομμυρίων. Όπως ξέρουμε είναι υποθετικό το νούμερο αυτό και όπως ξέρετε σε πολλές χώρες δεν θα υιοθετηθεί από αυτή την προγραμματική περίοδο και για τον Jaspers ε, ε, το Jaspers είναι μια κοινή κοινοπληξία. Συμμετέχουν ε, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Οικονομική ανάπτυξη ε, και, και KW και θέλουμε να παράσχουμε τεχνική βοήθεια στα νέα κράτη-μέλη. Η τεχνική αυτή βοήθεια παρέχεται στις δημόσιες αρχές που αναλαμβάνουν να προετοιμάσουν ε, μεγάλα επενδυτικά προγράμματα. Η βοήθεια που δίνεται είναι στήριξη με εμπειρογνώμονες, δηλαδή Εργαζόμαστε με έναν τρόπο έτσι ώστε να συμμετέχουν οι εμπειρογνώμονε στην προετοιμασία μεμονωμένων προγραμμάτων είτε να παράσχουν οριζόντιου χαρακτήρα συμβουλέ, Δηλαδή όταν προετοιμάζουν μια στρατηγική σε ένα συγκεκριμένο τομέα για ε, την ανάπτυξη συνδρομικού δικτύου λόγου χάρη ή όταν μιλάμε για συστήματα διαχείρισης λιμάτων κτλ. Δηλαδή παρέσχουν συμβουλές στην κυβέρνηση για να τους προετοιμάσουν γιατί το τελικό στόχος είναι να είναι σε θέση εγκαίρως να προετοιμάσουν μεγάλα προγράμματα και να τα υποβάλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και όπως ε, είπατε κι εσείς, ε, πτυχές της ποιότητας και της συμμόρφωσης με την κοινωτική νομοθεσία είναι αυτονόητο ότι όταν έχουμε να κάνουμε με περιβαλλοντικά project, ε, οι εμπειρογνώμονες θα παρέχουν συμβουλές για τις κύριες απαιτήσει που θα πρέπει να πληρούνται, τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να γίνει αποδεκτό τελικά το πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το σύστημα είναι στη διάθεση των κρατών μελών, αλλά έχει και αντίκτυπο. Δηλαδή, εμείς ενδιαφερόμαστε από την πλευρά της Κομισιόν να λαμβάνουμε προγράμματα καλής ποιότητας που θα παρουσιάζονται και ταχύτερα από τα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ πολύ, Ρούντολφ, και θα ήθελα εδώ να ολοκληρώσω τώρα τη συνεδρίαση. Θα συναντηθούμε σε μία εβδομάδα στις 9 Δεκεμβρίου 5 στις 9 το πρωί. Θέλω επίσης να σας παρακαλέσω να ε, μην αργήσετε γιατί έχουμε πολύ βαριά ημερήσια διάταξη. Θα σας αποφασίσω και για τις αποφάσεις των νηστών που πήραμε χθε και για το Στρασβούργο και για την ε, συνεδρίαση ε, των αρμόδιων ε, υπουργών για τις περιφέρειες. Εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ όλους για την ενεργή συμμετοχή σας.